Uh, Παρακαλώ να καθίσουμε. Καλώς ορίσατε. Θερμό καλώς όρισμα και δεν θέλω να κάνω λογοπαίγνια με τον καιρό που έχει έξω. Πρώτη φορά μετά τις δεκοπές σας βλέπω όλους μαυρισμένους, ξεκούραστους και έτοιμους για δουλειά. Έχουμε τη μεγαλύτερη αίθουσα του Κοινοβουλίου στη θέση μα σήμερα, αλλά η αίθουσα δυστυχώ δεν έχει παράθυρα και έτσι δεν μπορούμε να απολαύσουμε τον ωραίο ήλιο. Αλλά έστω. Καλωσορίζω και όλους όσοι μας παρακολουθούν από το διαδίκτυο. Να σας εξηγήσω καταρχάς γιατί έχουμε αυτή τη μεγάλη αίθουσα σήμερα. και να προχωρήσω κάποιες ανακοινώσεις, αλλά πρώτα θα πρέπει να εγκρίνουμε επισήμω στην ημερήσια διάταξη. Η ψηφοφορία για την έκβαση του τριμερούς διαλόγου για το νέο νομοθετικό πακέτο της κυρίας Ομανρούιτσεν θα αναβληθεί. Το πρέπει να σας πω, διότι μπορούμε να έχουμε επιβεβαιωμένη συμφωνία με την Ιρλανδική Προεδρία, αλλά όταν πήγε το θέμα στο Κορεπέρ, ήγηραν πολλά κράτη-μέλη θέματα σχετικά με τις αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου και τα κατά πόσο μπορεί να παρίσταται σε συνεδριάσεις ομάδα, της ομάδας των εμπειρογνωμόνων. Θέματα και επιτροπολογίας, τα οποία θα γνωρίζουν ασφαλώς όσοι έχουν εντωμεταξύ ασχοληθεί με την ε, επιτροπολογία. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε σε συνεννόηση με την Λιθουανική Προεδρία, αλλά προσπαθούμε το μεταξύ να επιλύσουμε το πρόβλημα και κάνουμε και τις σχετικές επαφές με τους συγητές και συγκρότες συγητές. Αυτό για να είστε ενήμεροι. Πάντως, η ουσία των όσων είχαμε συμφωνήσει έχει εγκριθεί και δυστυχώ αυτό είναι το Αχ, έχει κολλήσει το θέμα στην επιτροπολογία. Δέχεστε την ημερήσια διάταξη λοιπόν. Καλώ ευχαριστώ. Και υπενθυμίζω ότι προβλέπεται ψηφοφορία στις 4 παρα 10 μαζί με την έγκριση της πρότασης για τις νόσες προμήθειες, τις συμβάσεις προκατακτικές ε, παρατηρήσεις επίσης, αν μου επιτρέπετε, για τα θέματα που έχουμε ολοκληρώσει και τη δουλειά που έχουμε μπροστά μας. Την προηγούμενη εβδομάδα, 26 Αυγούστου, ε, έγινε μια πολύ επιτυχής επίσκεψη στην Ελλάδα, με πολύ καλή προσέλευση και σε του επίπεδο επαφές με την ελληνική κυβέρνηση. Συναντηθήκαμε και με τον Υπουργό Κώστα Χατζηδάκη, τον οποίο φαντάζομαι θα θυμάστε πολύ ως ε, δραστήριο συνάδελφο. Ήταν και πρόεδρος της Επιτροπής των Μεταφορών, αν δεν απατώμε, για μεγάλο διάστημα. Τώρα είναι αρμόδιος Υπουργός για θέματα ανάπτυξης, υποδομών, οικονομικής ανάπτυξης μεταφορών και τουρισμού. Πολύ μεγάλο χαρτοφυλάκιο. Μας μίλησε για τα σχέδια του για την ε, εισαγωγή μέτρων της εσωτερικής αγοράς και μεταρρυθμίσεις στην ευρωπαϊκή, στην ελληνική οικονομία. Θα αναλάβει εκείνο την Προεδρία του στο Συμβούλιο στα σχετικά θέματα κατά την ελληνική Προεδρία. Και είμαστε η πρώτη επιτροπή πρέπει να πω που επισκεφθήκαμε την Ελλάδα εν ώψη της ανάληψης της Προεδρίας τον Ιανουάριο που προσβλέπουν με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό οι Έλληνες. Και ξέρουμε ότι θα τους απασχολήσει πολύ. Είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση και στο, Ευρωπαϊκό, στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Η κυρία Στάιλερ δεν ξέρω αν ακόμα ασχολείται με το, επιτρο... με το περιοδικό Parliament, κοινοβούλιο, αλλά όποιοι το διαβάζετε θα δείτε και μια δική μου αξιολόγηση, μια σύντομη επισκόπηση αυτής της επίσκεψης, αν σας ενδιαφέρει. Και κάτι άλλο. Εν συντομία, έχουμε την επόμενη, τον επόμενο μήνα ορίσει τον εορτασμό της ενίας αγοράς και την ανάπτυξη από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διαλόγου και ε, ε, διαδικτυακά με, με βουλευτές της Επιτροπής μας. Η Γενική Διεύθυνση για την εσωτερική Αγορά ασφαλώς θα, θα έχει έρθει σε επαφή μαζί σας, αν δεν το έχει πράξει ακόμη θα το πράξει. Αλλά πάντως μου ζήτησε να σας ενημερώσω και να σας καλέσω να λάβετε μέρος και στο διάλογο με πολίτες που θα αναπτυχθεί ε, καλό θα βέβαια να συμμετάσχουμε στο δυνατόν περισσότεροι ευρωβουλευτές με θέματα διαφορετικά, με διαφορετική πολιτική προέλευση και εθνική ασφαλώς. Ε, παρακαλώ να το σημειώσετε λοιπόν. Και επίσης θα έχετε δει στα πρακτικά, ε, στο φάκελό σας τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Μαΐου και του Ιουνίου και ως ήθιστε Εάν δεν έχουν διατυπωθεί αντιρρήσεις μέχρι το συνεδρία σα θα θεωρηθεί ότι εγκρίθηκαν. Κάλυψε όλα τα θέματα νομίζω. Και ξεκινώ την ε, φθινοπορεινή αυτή συνεδρίαση με το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για το Λιανικό Εμπόριο προς όφελος όλων των παραγόντων Όλοι οι σκιώδεις πλήν του κυρίου Σαλβίνη είναι εδώ, η κυρία Κοράτσα Μπίλτ είναι εδώ, η κυρία Ριγκόια Πέρες είναι, ο κύριος Κύριε η κυρία Ρίλε, αποφαινόμενος, η κυρία Ρίμπιντερ, εκ μέρους Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αν δεν απατώμε. Θα σας δώσουμε και σας το λόγο όταν έρθει η ώρα για, για την έκθεση του κυρίου Ντελιόγκ τον οποίο και παρακαλώ να μας παρουσιάσει το σχέδιο εκθέσεως για να ακούσουμε μετά τους οικειώδες, στην Επιτροπή και όποιον άλλον συνάδελφο επιθυμεί να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ, Μάλκομ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος, ε, διότι φαντάζομαι ότι μπορούν να τη διαβάσουν την έκθεση όλοι. Θα κάνω κάποια σχόλια για ζητήματα που μπορούν να μπορούμε να εξετάσουμε εδώ. Πρωτού αρχίσω να σας πω ότι πάντοτε ήταν αδυναμία μου το λιανικό εμπόριο. Όχι μόνο λόγω της μεγάλης του σημασίας ε, για τις οικονομίες μας, λέει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι το 15% της απασχόλησης είναι στο λιανικό εμπόριο και το 11% του ΑΕΠ μας ε, στην Ευρώπη. Ε, αυτά οφείλονται στο λιανικό εμπόριο, οπότε έχει μεγάλη βαρύτητα, αλλά όχι μόνο γι' αυτό, διότι ε, από την εμπειρία τους όλοι ξέρουν ότι η αγορά αγαθών και υπηρεσιών, ε, πέρα από την ίδια την αγορά, σχετίζεται και με την κοινωνική αλληλεπίδραση. Υπάρχει μια κοινωνική διάσταση στις αγορές που κάνουμε. Δηλαδή μια πόλη χωρίς μαγαζιά λιανικής δεν είναι πόλη. Οπότε χάρηκα που μου επέτρεψε η Επιτροπή να αναλάβω το ρόλο του εισηγητή για το σχέδιο δράσης για το λιανικό εμπόριο Ήθελα να εκπονήσω μια έκθεση χρήσιμη για τον τομέα, ε, χάρη στην οποία ελπίζω να σημειωθεί η πρόοδος. Μέσα σε αυτή την έκθεση έχουμε πολλές ε, ε, πτυχές του ζητήματος, διότι δεν ασχολούμαι μόνο με αυτό το σχέδιο δράση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και με την πράσινη βίβλο για τις αθέμητες πρακτικές ανταγωνισμού στο B2B και στον εφοδιασμό της αλυσίδας τροφίμων. Οπότε είναι πολυδιάστατο το ζήτημα, βεβαίως είναι ελένδετα όλα αυτά τα θέματα. Σίγουρα ε, κάποιοι συνάδελφοί μου θα απογοητευτούν, ε, διότι είναι ε, υπερβολικά σύντομες οι παράγραφοι, αλλά προσπάθησα να βάλω όσα περισσότερα ζητήματα μπορούσα μέσα στην έκθεση, κόμματα για τη δημιουργία της πραγματικής ενίας αγοράς για το λιανικό εμπόριο, για τις κοινωνικές πτυχές, την πτυχή της απασχόλησης, για τη βιωσιμότητα, ενδεχομένως να επιθυμούσατε να δείτε περισσότερα πράγματα σε σχέση με το τωρινό περιεχόμενο της έκθεσης. Απλώς ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι ευπρόσδεκτες είναι οι προσθήκες που θα προτείνετε και εγώ ίδιος υπομορφή τροπολογιών προς την ίδια μου την έκθεση θα εισηγηθώ προσθήκες, αλλά έχουμε περιορισμένο χώρο και ούτω ή άλλως ε, υπερεύει τα όρια χάρη στη γραμματεία και κατάφερα να χώσω και άλλα πράγματα μέσα. Ε, κάτι πολύ σημαντικό είναι ότι πρέπει να επικρατήσει ένας πλουραλισμός ε, πολυμορφίας στο λιανικό εμπόριο. Δηλαδή, δεν πρέπει να ασχολούμαστε μόνο με τις μεγάλες υπεραγορές, ε, τα μεγάλα καταστήματα λιανικής, αλλά και τα μικρότερα. Δεν πρέπει να πιστεύουν ε, ε, κάποιοι, α, ξέρω εγώ, εγώ δεν πηγαίνω ποτέ σε μεγάλα καταστήματα, δεν μ' αρέσουν, διότι από κοινωνικοπολιτισμική σκοπιά είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει ποικιλομορφία ε, στο, ως προς το μέγεθος των καταστημάτων και τα προϊόντα που προσφέρουν. Δηλαδή και τα ίδια τα καταστήματα θεωρούν ότι πολλούν περισσότερα αγαθά όταν ε, υπάρχει μεγάλη ποικιλομορφία σε, ένα, ε, σε μια περιοχή όπου υπάρχουν καταστήματα, σε μια εμπορική περιοχή, γιατί έρχονται περισσότεροι άνθρωποι και στη Γαλλία και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το ίδιο έχει διαπιστωθεί ότι Βλέπουμε λοιπόν ότι με αυτό το μίξ που γίνεται, με την ποικιλία που υπάρχει, έχουν ε, καλύτερα αποτελέσματα στην ε, οικονομική τους χρήση στα καταστήματα. Αν εξετάσουμε την ε, τωρινή κατάσταση και την οικονομική κρίση, ε, τα μικρότερα καταστήματα υφίστανται τις ε, σοβαρότερες απειλές και εν γένει. Αν συγκρίνω την έκθεσή μου με το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όντως προσδίδω εγώ πολύ μεγαλύτερη σημασία στο θέμα της κρίσης που βιώνουμε, διότι αυτά μου λένε οι ότι αυτή είναι η προτεραιότητά μας. Ε, και βλέπουμε ότι η εμπιστοσύνη των καταναλωτών ευθύνει σε πάρα πολλές χώρες ε, ίσως ε, δεν είναι αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά σίγουρα με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Διακυβέρνηση και το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο έχει μεγαλύτερες δυνατότητες η Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν με αντιστάθηκα στον πειρασμό να κάνω και μία αναφορά στο γιατί τα κράτη-μέλη, κάποια κράτη-μέλη συνεχίζουν να αυξάνουν ε, τη φορολόγηση για το λιανικό εμπόριο, κυρίω ε, μιλώντα για το ΦΠΑ. Το βλέπω στην Ολλανδία, στη χώρα μου, αυξήθηκε κατά δύο ποσοστίε μονάδε το ΦΠΑ και ε, αυτόματα σημειώθηκε πτώση στι πωλήσει του λιανικού εμπορίου και η εμπιστοσύνη των καταναλωτών είναι σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, εξακολουθεί να είναι μάλλον σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα στη χώρα μου. Με αυτά λοιπόν πιστεύω ότι πρέπει να σκεφτούν σοβαρά τα κράτη-μέλη περαιτέρω αυξήσει του ΦΠΑ που πλήττουν ε, τον τομέα του λιανικού εμπορίου. Δεύτερον, είμαι πεπισμένο πως ε, οι επιχειρηματίες ε, δύναται να βρουν δικές τους λύσεις για αυτό το πλήθος προκλήσεων που αντιμετωπίζουν ταυτόχρονα. Βλέπω πολλαπλά παραδείγματα και στην Αγγλία και στη χώρα μου ε, δημοσίων πολιτικών με στόχο να ζωγονηθούν οι βασικοί εμπορικοί δρόμοι, να γίνουν νέοι σχεδιασμοί ε, και να υποδείξουν τι είδους καταστήματα επιθυμούν, δηλαδή καινοτόμα καταστήματα, ε, που προσπαθούν να προσελκύσουν στις εμπορικές περιοχές των πόλεων. Και αυτό που θέλησα να κάνω είναι μέσω της έκθεσης να συνειδητοποιήσω αν συμφωνεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι χρειάζεται περισσότερη ευελιξία σε σχέση με του κανόνε ανταγωνισμού ή του κανόνε για την εγκατάσταση νέων καταστημάτων. Δεν είναι μια οικονομική πολιτική, δεν πρέπει να είμαστε προστατευτικοί. Είναι μια πολιτική ε, που στόχο έχει κάποιε γειτονιέ, κάποιε συνοικίε ε, να να παραμείνουν γνωστές ε, ως ε, εμπορικές ε, περιοχές. Ε, αυτός δεν είναι ο ρόλος του επιχειρηματία, διότι ο επιχειρηματίας ασχολείται με την επιχείρησή του να αντιστήσει να την Πρόκειται πλέον για χωροταξικό σχεδιασμό και αν δούμε τις άδειε πολεοδομίας, οι τοπικές αρχές σίγουρα μπορούν να δώσουν κάποιες κατευθύνσεις ή να υποδείξουν τη σωστή κατεύθυνση μέσα από τα μέτρα που επιβάλλουν. Ως προς την προστασία των μικρών καταστημάτων, ε, σε σχέση με τα περιτά ε, προσκόμματα που υπάρχουν στην ενιαία αγορά και προστασία από κυβερνητικές ρυθμίσεις που δυσκολεύουν περισσότερο τη ζωή των επιχειρηματίων. Ε, το αναφέρω και αυτό στην εκθεσή μου. Κάτι άλλο τώρα που παρατήρησε και ίσως δημιουργήσει σύγχυση. Το θέμα του ηλεκτρονικού εμπορίου. Δεν είμαι καθόλου κατά του ηλεκτρονικού εμπορίου. Το αντίθετο είναι απαραίτητο ε, και είναι μια εξέλιξη ακόμη και αν εδώ στην Επιτροπή που με δεν μας αρέσει δεν έχει καμία σημασία γιατί το ή άλλως θα, εδώ είναι, θα παραμείνει και θα αναπτυχθεί και δημιουργεί πλήθο ε, πλήθος νέων ευκαιριών ακόμη και στο λιανικό εμπόριο. Δεν πρέπει να το εκλαμβάνουμε ως απειλή αλλά ως ευκαιρία. Ε, θέλησα όμως να τονίσω ότι για ε, τα μικρά ανεξάρτητα καταστήματα συνιστά και μεγάλη πρόκληση. Μίλησα με πολλούς ε, μικρού καταστηματάρχε που μου είπαν ε, ότι είναι κατάστηματάρχε. Θέλουν να έχουν το κατάστημα και να βλέπουν ανθρώπου. Δεν θέλουν να γίνουν γραμματοθυρίδα ηλεκτρονική. Θέλουν επαφή. Υπάρχουν ε, κάποιες, ε, θα έλεγα, παράλογες αντιρρήσεις, όμως πρέπει να τις εξετάσουμε. Δηλαδή, αν πούμε, αν το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι σημαντικό για σας, δεν θα αλλάξει τίποτα. Με κάποιο είδους πολιτική θα βρούμε μια ε, πολύμορφη πολιτική που θα ταιριάζει και στους μικρούς καταστηματάρχες. Ε, δηλαδή, τους πρότεινα εγώ, γιατί δεν φτιάχνετε κι άλλη μια ιστοσελίδα. Δηλαδή, θα υπάρχει σχέση ανάμεσα στο κατάστημά σας και την ιστοσελίδα σας. Σταδιακά γίνεται αυτό αντιλήπτο, αλλά θέλει προσπάθεια. Αν δεν γίνει όμως αυτό, ε, θα ε, χάσει το τρένο το μικρό κατάστημα, θα χάσει τις εξελίξεις ε, του ψηφιακού εμπορίου και θα χάσει έδαφος στην αγορά και μερίδιο στην αγορά. Δηλαδή, ε, Στι συζητήσει μας για το ηλεκτρονικό εμπόριο δεν αναφέρομαι συχνά σε αυτό το ζήτημα και γι' αυτό νιώσα την ανάγκη να το τονίσω. Για το franchising επίση ε, είναι ένα άλλο ζήτημα που πρέπει να εξετάσουμε. Δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες. Δεν λειτουργούν όλα ε, ομαλά Όπω έχει τώρα η κατάσταση, θα πρέπει να προσέξουμε. Το δεύτερο τμήμα τώρα. Αθέμητε εμπορικέ πρακτικέ. σε κάποιους κύκλους θεωρείται ως μια κίνηση κατά των αναπτυσσομένων χωρών, ε, του περιβάλλοντος και των ε, γεωργών πιο συγκεκριμένα. Δεν μπορώ να δεχτώ αυτές τις κατηγορίες. Ε, Θα άλλαζε και πολιτική οικογένεια, μα ήταν έτσι. Αλλά μέσα από τις διαβουλεύσεις ε, και πολλαπλές συνομιλίες, ε, ακόμη και με ενώσεις ε, παραγωγών κτλ. Προσπάθησα να καταλάβω ποιο είναι ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπίσουμε αυτές τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές. Και εν κατακλείδη δεν είμαι πεπισμένος ότι η νομοθεσία είναι η βέλτιστη λύση για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Αν θεσπίσουμε νέα νομοθεσία για τις αθέμητες πρακτικές, σίγουρα θα υπάρχουν παραθυράκια και κάποιες εταιρείε μπορεί να υποχρεωθούν να ε, επιχειρήσουν ε, να χρησιμοποιήσουν αυτά τα παραθύρα και να παρακάμψουν την ομοθεσία Δεν είναι ο αποτελεσματικότερος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα προς το παρόν ταυτόχρονα. Ε, υπάρχει η εθελοντική πρωτοβουλία του τομέα, όπως ονομάζεται. Στις 16 Σεπτεμβρίου θα ε, δρομολογηθεί επίσημα, θα ανασαριστεί επίσημα. Ε, και όλοι οι εμπλεκόμενοι, όχι μόνο τα σούπερ μάρκετ και η παραγωγή, αλλά και οι ενδιάμεση, μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν πολλοί ε, παραγωγοί και διανεμητές ε, που παίρνουν πολύ μεγάλο ποσοστό του κέρδους. Δεν είναι υπεραγορές, αλλά είναι διάμεση ανάμεσα σε εταιρείε δηλαδή και προσπαθούν εκείνοι να βρουν τη λύση και να την εφαρμόσουν. Ας τους δώσουμε την ευκαιρία τους ε, να δείξουν ότι είναι μια σοβαρή πρωτοβουλία και να δούμε αν μπορεί στην πράξη να λειτουργήσει. Αν όλοι υιοθετήσουν αυτή τη λύση και υπάρχει βούληση στον τομέα να εφαρμοστεί, σίγουρα θα είναι πολύ πιο αποτελεσματικό από ότι ένα επιπλέον νομοθέτημα πρέπει να εφαρμοστεί και ξέρουμε όλοι ποια προβλήματα υπάρχουν, οι καθυστερήσει, πόση προσπάθεια μα χρειάζεται για να το καταφέρουμε, αν είναι τελικά αποτελεσματικό κτλ. Ε, έχω κάποιες συστάσεις, αλλά και για την ίδια το, η πρωτοβουλία. Αν το θέμα της εφαρμογής, προτείνονται κάποιοι μηχανισμοί, αλλά ουσιαστικά βάσει της πρωτοβουλίας χρησιμοποιούνται οι φυστάμενοι εθνικοί μηχανισμοί ε, και αυτοί οι μηχανισμοί θα χρησιμοποιηθούν για να ε, ρυθμιστούν νομικές διαφορές. Κάποιες εταιρείες περιμένουν Μάλλον δεν θα, πρέπει να περιμένουμε μήνες και χρόνια ε, για να δούμε αν θα λειτουργήσει αυτή η λύση, γιατί αν Βεβαίως ε, σε αυτή την ε, περίπτωση ίσως προσχωρήσουν και άλλες ενώσεις παραγωγών σε αυτή την πρωτοβουλία. Δεν νομίζω ότι υπονομεύεται έτσι η πρωτοβουλία. Τους δίνουμε μια ευκαιρία για να δούμε αν θα λειτουργήσει στην πράξη. Αυτή είναι η πρώτη μου σύσταση. Η δεύτερη σύσταση που κάνω είναι να αποστασιοποιηθούμε από κάποιες εθνικές δράσεις κάποιων κρατών μελών πώληση κάτω της τιμής του κόστους. Τιμής που πλήρωσε δηλαδή το σούπερ μάρκετ για τα τρόφιμα παραδείγματος χάρη. Νομίζω μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι θα επικρατήσει ένα σύστημα που θα απαγορεύει τέτοια πρακτική και θα δίνει μια εγγύηση. Μίλησα με εκπροσώπους ε, μεγάλων σούπερ μάρκετ που συμφώνησαν ε, ατύπως με αυτή τη λύση. Δημιουργεί ένα χώρο μίσου όρου ανταγωνισμού ουσιαστικά και πολλά σούπερ μάρκετ θα χαίρονταν αν δεν χρειαζόταν να ανταγωνιστούν και να πολλούν ε, κάτω από το κόστος για να παραμένουν ε, ανταγωνιστικά. Θα κλείσω τώρα και φυσικά με στη διάθεσή σας, μπορούμε να επανέλθουμε. Μάλιστα, πολύ ωραία. Έχουμε 20 με 25 λεπτά στη διάθεσή μας να ακούσουμε τα σχόλια των σκιωδών και οποιοδήποτε άλλο συναδέλφου θέλει τον λόγο. Στάιλερ είναι ήδη στον κατάλογο, κάποιος άλλος. Παρακαλώ σηκώντε τα χέρια σας να σας ε, εγγράψω στον κατάλογο. Ε, κύριε Κοράτσα Μπίλ θα πάρει πρώτα το λόγο γιατί είναι η συγγήτρια εκ μέρους του ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να καλωσορίσω θερμά ο συναδέλφος και να ευχαριστήσω τον Κορνέλιους για την πολύ καλή δουλειά που έχει κάνει. Συμφωνούμε με το μεγαλύτερο μέρος των προτάσεών του και αυτό ε, δείχνει και ότι και η Κομισιόν και το Κοινοβούλιο εργάζονται ε, σε μια νέα προοπτική. Υπάρχει συνέχεια στο έργο μας. Είχα και εγώ κάνει μια έκθεση ε, για την αγορά στην Ευρώπη το 2011 την εγκρίναμε, συγκεκριμένα για το λιανικό εμπόριο. Ε, θέλαμε να εγγραφεί στο πολιτικό χάρτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στο επίπεδο που του αξίζει. Και επίσης αναγνωρίζουμε τις λιανικές πωλήσεις, το λιανικό εμπόριο, τη σημασία τους και θέλουμε η κρίση να μην επηρεάσει τις πάρα πολύ θεαματικές δυνατότητες απασχολησιμότητας που δείχνει ο τομέας αυτός που αποδεικνύεται ανθεκτικός ακόμα και στην περίοδο της κρίσης. Με το σχέδιο δράση ελπίζω να καταφέραμε να υιοθετήσουμε μια ρεαλιστική προσέγγιση για να δούμε συγκεκριμένα πώς μπορούμε την ελευθερία και τη δικαιοσύνη να τις εξασφαλίσουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και στις απομονωμένες περιφέρειες να υπάρχει πρόσβαση ε, σε ελεύθερες επιλογές, διαφοροποιημένες επιλογές ε, για τους καταναλωτές. Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να το πετύχουμε αυτό να προστατεύσουμε, αλλά ανοίγοντας ε, την αγορά, να στηρίξουμε την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία, τα είπε και ο Ντένις, και να φροντίσουμε ότι ε, μπορούν να είναι ανταγωνιστικοί. Δεν μπορούμε με δημόσιες παρεμβάσεις ε, και με επιδοτήσεις να προχωρούμε. Αν αυξάνουμε το δημόσιο, το κρατικό χρέος και σε εθνικό και στοπικό επίπεδο, δεν θα εξέλθουμε ποτέ από την κρίση. Μου άρεσε πολύ Ντένις λοιπόν που επέμεινε ότι δεν θα πρέπει να είμαστε προστατευτικοί, να ακολουθήσουμε πρακτικές προστατευτισμού και ελπίζω να εμείνει σε αυτή τη γραμμή. Θα ήθελα επίσης να πω ότι ε, οι δοκιμές, ε, η εξέταση οικονομικών αναγκών είναι ένα θέμα σημαντικό. Ήμουν εισηγήτρια και για την έκθεση περί υπηρεσιών. Το ίδιο πρόβλημα είναι, διότι οι οικονομικές ανάγκες ουσιαστικά εξισώνεται με τον αμυγή προστατευτισμό. Δημιουργεί προβλήματα, περιορίζεται την ελευθερία κυκλοφορία αγαθών ε, και την ελευθερία εγκατάστασης. Θα κάνω τροπολογίες, σας ε, το λέω ευθύς εξ αρχής, Επίσης, αυτή η διόρθωση και η διευκρίνηση που έκανε στην οποία εκτιμώ ιδιαίτερο για το πώς βλέπεις το ηλεκτρονικό εμπόριο, επίσης μας βοηθά πολύ. Δεν είναι απειλή, είναι ευκαιρία, είναι συμπλήρωμα. Ε, κάποιοι το φοβούνται, δεν μπορούμε όμως να το σταματήσουμε, είναι μια θετική εξέλιξη. Σίγουρα λοιπόν θα πρέπει να διευκολυνθεί και να ενθαρρυνθεί σε ό,τι αφορά το B2B, business to business. Πάλι είμαστε στο μικρό σχήμα. Ε, πέρασε ο καιρό ε, για να είμαστε ιδεολόγοι απλά. Πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα ρεαλιστικά. Ούτε τίθεται θέμα να τιμωρηθούν οι ισχυροί ή να θυματοποιηθούν οι μικρότεροι. Το θέμα είναι να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια, μεγαλύτερη δικαιοσύνη. Και αυτό αποδίδει όχι μόνο στις Βρυξέλλες, αλλά στην πραγματική ζωή, στις χώρες μας. Το βλέπουμε ελευθερία επιλογής, ε, ε, να έχει αξία, ε, να είναι αποδοτικές υπηρεσίες που παρέχουμε, να υπάρχει το value for money και πρέπει να συγχαρούμε τα μέλη της πλατφόρμας που ενέκριναν όχι μόνο τις αρχές αλλά και τα εκτελεστικά εφαρμοστικά μέτρα. Θα έχουμε την υπογραφή από πολλούς ελπίζουμε πρωταγωνιστές και ελπίζουμε και οργάνωση των αγροτών που πάρα πολύ ενεργά και επιδομητικά συμμετείχαν σε όλη τη διαδικασία. Ελπίζουμε να ε, ληφθούν υπόψη και των δικών τους οι απόλυτα θεμητές ανησυχίες ώστε να είναι όλοι ικανοποιημένοι. Με την βοήθεια λοιπόν της Κομισιόν και με την πίεση που ασκεί, με την μελέτη εξολόγηση επιπτώσεων και τις άλλες τις μελέτες θα έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Αυτό που είναι σημαντικό αυτή τη στιγμή κατά την άποψή μου είναι ουσιαστικά να ελέγξουμε τα αποτελέσματα και να μην ε, μιλάμε θεωρητικά. Ε, πρέπει να δώσουμε σάρκα και οστά ε, σε αυτές τις προτάσεις και οι δίκαιες πρακτικές να ισχύσουν στην πράξη, να δούμε μια αλλαγή νοοτροπίας. Επίσης, σε ό,τι αφορά τη βιωσιμότητα, Ντένι ξεστηρίζω, είναι πολύ σημαντικό οι λιανέμποροι και οι να αναλάβουν την ευθύνη τους, Όπω και πράττουν άλλωστε. Υπάρχουν σειρά θελοντικών μέτρων, υπάρχει επένδυση στην καινοτομία, στην έρευνα και την ανάπτυξη, σε μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση. Αυτά πρέπει να συστούν. Επίση, στηρίζω τον τέννις και στο θέμα τη ετικετοθεσία, της επισήμανσης διότι βλέπουμε να υπάρχουν όλο και να πλαπλασιάζονται διάφορες προτάσεις και κάτι τέτοιο δεν ωφελεί τον καταναλωτή, δεν είναι σαφές το τοπίο. Θα συνεργαστώ με τον συγκεκριτή και του Σκιώδης, θα προσπαθήσω να μην χάνουμε ε, από το μυαλό μας τη σημασία που έχει το τομέας του λιανεμπορίου και έχουμε και τον πρώτο γύρο, ε, το πρώτο τραπέζι αν θέλετε, πρώτο γύρο συζητήσεων ε, για ένα δίκαιο αποτελεσματικό λιανικό εμπόριο στην Ευρώπη. Εκεί η πλευρά της προσφοράς, η πλευρά των λιανεμπόρων θα μπορέσει να μας παρουσιάσει την κατάσταση, να εκθέσει τα θετικά, τα αρνητικά, το B2B, business to business και για μας νομίζω ε, είναι πολύ καλή ε, χρονική στιγμή για να στηρίξουμε τους ε, λιανεμπόρους, για να δώσουμε θέσεις εργασίας στην Ευρώπη. Πρόεδρος, ναι, θα το έλεγα κι εγώ, αλλά το είπες πάρα πολύ εύγλωτα. Επαναλαμβάνω λοιπόν για όποιον θέλει να το παρακολουθήσετε. Θα είναι στις 26 Σεπτεμβρίου στις 3 αυτή η εκδήλωση. και όποιος θέλει ε, είτε από την πλευρά των ελληνικών είτε από την πλευρά των προμηθευτών μπορεί να μας συναντήσει στις 26 Σεπτεμβρίου και να παρακολουθήσει. Κύριε Ριγκόγεν Πέρφ, τώρα έχει το λόγο από την πλευρά των Σοσιαλδημοκρατών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα εκφράζω την ικανοποίησή μου για την πολύ καλή έκθεση του κυρίου Ντεγιόν και είναι ένα κείμενο που θεωρώ ότι είναι άρτιο ισορροπημένο και συμφωνώ σχεδόν ε, στο σύνολο, με το σύνολο των προτάσεων. Όπως ε, τονίζεται στην έκθεση, όλοι γνωρίζουμε ότι το λιανεμπόριο είναι πάρα πολύ ε, σημαντικό στο μέσα στην ανάπτυξη και της παραγωγικότητας και την ανάπτυξη και υπάρχουν ε, μοντέλα πιο ε, βιώσιμα τα οποία θα πρέπει να προαχθούν. Όμως η οικονομική κρίση, οι πολιτικές λιτότητας επηρεάζουν, πλήττουν ε, τον τομέα αυτό άμεσα. Βλέπουμε συνεχή υποχώρηση των πωλήσεων και συνεχές πτώσεις στις τιμές στα στοιχεία. Και αυτό δείχνει ότι μειώνονται σε όλους τους τρόπους, σε όλες τις μορφές διανομής ε, το λιανικό εμπόριο. Και αυτό βέβαια επηρεάζει πιο πολύ τους ανεξάρτητους, ε, τους αυτοαπασχολούμενους και τις μικρές αλυσίδες. Ο κ. Δεγιόγκ είπε ότι ε, μια πόλη χωρί καταστήματα είναι νεκρή πόλη. Αυτό για το οποίο μιλάμε δεν είναι προστατευτισμός. Θέλουμε να υπάρχει ισορροπία. Ε, να επιβιώνουν ε, οι μικρές, μεσές και μεγάλες επιχειρήσεις και τα σούπερ μάρκετ αλλά και οι οικογενειακέ επιχειρήσει. Όπω στη χώρα μου έπεσε 10,6% το λιανεμπόρ και στα στις αλυσίδες αυτές βλέπουμε πάρα πολύ και συνεχή και διαρκή μείωση του κύκλου εργασιών. Πιστεύω ότι θα πρέπει μεταξύ άλλων να δούμε και κάτι άλλο. Πρώτα απ' όλα πώς επηρεάζει η οικονομική κρίση τον κλάδο αύξηση του ΦΠΑ, των συντελεστών, ε, επανακατατάξεις ε, προϊόντων, ε, πρόβλημα με τις πιστώσεις, τις χορηγήσεις, επίσης εργασιακές σχέσεις, καταχρήσεις στο λιανικό εμπόριο. Κάτι το οποίο πλήττει κυρίως τις γυναίκες, τους ανειδίκευτους ανθρώπους με χαμηλή δίκευση και τους μετανάστες. Επίσης, κατά πολέμηση της παραοικονομίας, ε, της φοροδιαφυγής, ε, υποφυγή γραφειοκρατικών εμποδίων που καθυστερούν ε, τον χρόνο για το άνοιγμα ενός καταστήματος. Επίσης, μεταγκατάσταση των επιχειρήσεων διανομής και προμηθειών, οι οποίοι εκμεταλλεύονται πιο χαλαρές νομοθεσίες. Βέβαια χρειάζονται να δούμε και άλλα θέματα, την, πώς θα προωθήσουμε τις τοπικές αγορές, ε, το εμπόριο, πώς θα ε, άρουμε διοικητικά εμπόρια, πώς θα αποφύγουμε την κανονιστική διασπορά, την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, πώς θα προωθήσουμε το χωροτεξικό σχεδιασμό, πώς θα διατηρήσουμε την ιστορική και καλλιτεχνική κληρονομιά. Με ικανοποίηση βλέπω ότι υπάρχει αυτή η θελοντική πρωτοβουλία και αυτό είναι ένα πρώτο βήμα. Νομίζω όμως ότι θα πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι σε αυτό το θέμα, διότι οι, εμπορικές, οι αθέμητες εμπορικές πρακτικές είναι ένα από τα βασικά εμπόδια που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Το λιανικό εμπόριο πρέπει να ε, το προστατεύσουμε από τις καταχρήσεις και πρέπει να επιδείξουν και κοινωνική ευαισθησία. Όλα αυτά είναι πολύ απαραίτητα για να βελτιωθεί η παραγωγικότητα. Τέλος, να ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά τον εισηγητή της έκθεση ε, και να σας ε, πω ότι και εγώ θα υποβάλω τροπολογίες με βάση όσα σας δήλωσα. Ευχαριστώ. Uh, thank you very much. Uh, Mr. Ευχαριστώ. κύριε Λόχεγκάρτ. Παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ καταρχάς για την παρουσίαση. Η έκθεση είναι πολύ καλή. Εμπεριστατωμένη. Κύριος Τεγιόγκ, ασφαλώς, έχει επιληφθεί κάποιον από τα πιο σημαντικά θέματα. Με ανησυχεί και για τη δική μου πατρίδα η κατάσταση στον τομέα του λιανικού εμπορίου. Θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις ε, συνέπειες της κρίσης. Υπάρχει βέβαια συζήτηση ιδιαίτερα για τα μικρά καταστήματα στο κέντρο των πόλεων. Δεν νομίζω να αμφισβητεί κανείς ότι κάτι πρέπει να γίνει. Διαφωνία προς τις μεθόδους που θα χρησιμοποιήσουμε μπορεί να υπάρχει. Και εμείς ε, τήρουμε να συμφωνήσουμε την κυρία Κοράτσα Μπίλτ. Ότι δηλαδή δεν είναι λύση ο προστατευτισμός, ότι πρέπει να έχουμε στο δυνατόν πιο ανοιχτή αγορά. Ε, βέβαια, ακούστηκε και η θέση ότι δεν ε, είναι ο προστατευτισμός το ζητούμενο. Χαίρομαι γι' αυτό, πολύ καλή αρχή. Θα πρέπει όμως και στην πράξη να δούμε τι σημαίνει. Και οι φιλελεύθεροι θα ακολουθήσουν κάθε καλή πρόταση στο βαθμό που δεν συνεπάγεται παρεμβατική πολιτική από το κράτος. Κάποιες γενικές παρατηρήσεις για τις κατευθυντικές μας γραμμές, τους φιλελευθέρους. Ε, στόχος λοιπόν η διαφάνεια, αποτελεσματική εφαρμογή και χρήση της φυστάμενης νομοθεσίας, όπως ακούστηκε στην καλή αυτή ακρόαση που έγινε χτες, πολλά είναι τα προβλήματα. Διαφαίνεται τάση προστατευτισμού στον τομέα αυτών που όμως δεν δίνει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Μια αποτελεσματική λοιπόν εφαρμογή είναι σημαντική. Θα καταθέσουμε τις σχετικές τροπολογίες. Η εξασφάλιση ενός περιβάλλοντος το οποίο να μπορεί να ανθίσει το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι επίσης ζητούμενο. Βλέπω ότι αναφέρεται στο ηλεκτρονικό εμπόριο και ο εισηγητής. Με μεγάλη ικανοποίηση σημειώνω ότι δεν τάσεστε εναντίον του. Χωρίς βέβαια να περίμενα κάτι τέτοιο, ήθελα να το επισημάνω. Το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι ο δρόμος για το μέλλον. Και πιστεύω ότι θα πρέπει και ο ίδιος ο τομέας να αντιληφθεί ότι ειδικά οι μικροί, τα μικρά ε, καταστήματα λιανικής θα πρέπει να ξεπεράσουν αυτόν τον πολιτισμικό φραγμό. Ξέρω ότι για τους πιο μεγάλους από εμάς στην ηλικία, από εμάς στην ηλικία είναι ίσως δύσκολο να το αναλογιστούν, αλλά μπορούν χωρίς ε, να χρειαστεί να βάλουν λουκέτο στο κατάστημά τους, να στραφούν στο, ηλεκτρονικό εμπόριο. Και αν καταφέρουμε ένα πλαίσιο μαζί με τον τομέα αυτό, νομίζω ότι μπορούμε να δώσουμε καλές λύσεις. Νομοθεσία. Αναμφίβολα είναι σημαντικό για την ε, απασχόληση και την ανάπτυξη στην Ευρώπη. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε λοιπόν για να επιτρέψουμε στον, στο λιανικό εμπόριο να αναπτύξει το δυναμικό του. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να δημιουργήσουμε το πλαίσιο αυτό για το μέλλον και αυτό συνεπάγεται βέβαια και ένα βαθμό νομοθετικής παρέμβασης που όμως θα πρέπει τα νομοθετήματα αυτά, όποια είναι, να γίνονται και σεβαστά με τις συνέπειες που αυτό μπορεί να έχει για ένα κράτος μέλος το οποίο ενδεχομένω δεν τηρεί τις σχετικές δεσμεύσεις. Είναι ένα θέμα το οποίο έχουμε συζητήσει πολλές φορές, χρόνια τώρα το ζητάμε. Έχει έρθει η ώρα τώρα νομίζω να κάνουμε κάτι. Και σταματώ εδώ. Έχω βέβαια σχόλια για πολλές από τις παραγράφους, αλλά δεν μου επιτρέπει ο χρόνος μου. Σταματώ λοιπόν εδώ και περιμένω να ακούσω και, προσβλέπω στη συνεργασία με τους, με τους συναδέλφους. Πρόεδρος, ναι βεβαίω. θα συνεχιστεί η συζήτηση. Κυρία Ρούλε, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη, γιατί περνάει η ώρα. Θα ήθελα να ευχαριστώ τον κύριο και είναι πολύ καλή η εξισορρόπηση του, του κειμένου του και σε αυτό θέλω να, υπογραμ... να επιμείνω γιατί δεν πρέπει να λησμονούμε ότι πρόκειται για ένα από του πιο διαφιλονικούμενους, για του πιο αμφισβητούμενου τομεί. Τις τελευταίες ώρες και ημέρες τις πέρασα στο γραφείο μου ε, δεχόμενοι πάρα πολλά τηλεφωνήματα, είτε εγώ προσωπικό είτε οι συνεργάτε μου, που ε, προσπαθούσαν να ανατρέψουν τις ισορροπίες. Αυτό που βλέπω εγώ στην έκθεση είναι ότι διατηρεί μια πολύ λεπτή ισορροπία και θεωρώ ότι δεν πρέπει να κατατεθούν τροπολογίες για να μην ανατραπεί ακριβώς αυτή η ισορροπία. Θα ήθελα να αναφερθώ ιδιαίτερα στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δράσης για την ε, ε, και τη δυνατότητα συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων. συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων είναι η πιο σημαντική διάσταση στην υπόθεση αυτή με την κυρία Κοράτσα Μπίλτα και με την προηγούμενη έκθεση είχαμε έρθει σε αντιπαράθεση γιατί υπάρχουν δυνατότητες και ε, αντιπαράθεσης μεταξύ των εμπόρων, μεγάλων, μικρών, στον ίδιο τομέα του εμπορίου, σε άλλο τομέα, εσωτερικό, εξωτερικό, γεωργία, ε, μεταποιημένα προϊόντα. Ε, εν πάση περιπτώσει είναι άπειρα τα προβλήματα που μπορεί να ανακύψουν και δεν πρέπει να λησμονούμε ποιες είναι οι προοπτικές για το μέλλον αυτού του τομέα μέσα στα πλαίσια της μεγάλης οικονομικής κρίσης που διανύουμε. Είναι πολύ καλό το κείμενο του κυρίου Ντεϊόγκ. τον ευχαριστώ θερμά. Και αναγνωρίζω ότι μπορεί ορισμένοι να θεωρήσουν στο σημείο 9, ναι μάλλον στο 9 πάνω απ' όλα, ε, δύσκολο να δεχθούν το, την αναφορά στις τοπικές αρχές ε, δημοτικές αρχές και τη δυνατότητα για αυτές να αναλάβουν δράση και προγραμματισμό. Ξέρω ότι ο προγραμματισμός ε, μπορεί να ακούγεται κάπως ε, δίσπεπτος για ορισμένους, αλλά δεν μπορούμε να τον παραγνωρίσουμε ως πάρα πολύ σοβαρή και σημαντική δυνατότητα να στηρίξουμε το λιανικό εμπόριο. Και πιστεύω ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε μια επιτυχή διασύνδεση μικρών και μεγάλων καταστημάτων και στα εμπορικά κέντρα να έχουμε ένα καλό μείγμα και από μεγάλα και από μικρότερα ε, καταστήματα. Γι' αυτό χρειάζεται προγραμματισμός. Ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Πολύ σύντομα και εγώ, ως Σκιώδης, στο ίδιο θέμα. Ξέρετε ότι με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Και ευχαριστώντας και τον κύριο Ιόγκ και όλους τους συναδέλφους που έχουν ασχοληθεί με το θέμα. γιατί ξέρετε ότι είναι πολλοί οι τομεί στο εμπόριο και όχι μόνο το εμπόριο τροφίμων που έχουν ιδιαίτερη σημασία. Σα ευχαριστώ λοιπόν όλου όσοι εργαστήκατε ενθουσιαδό για το θέμα αυτό. Μέσα στο περιορισμένο ρυθμό λέξεων μια εκθέσεω, κύριε Τελειώνη, νομίζω ότι καταφέρατε να κάνετε πάρα πολύ καλά πράγματα. Δύο-τρία πράγματα μου θέλω να υπογράψω από πλευρά μου. Καταρχάς, στην αγορά των αγαθών, δεν θέλω να επισημάνω για όσοι έχουν παρακολουθήσει το θέμα της σχετικής οδηγίας, ότι οι διαφορές ε, σε τιμές, ακόμη και για σχετικά βασικά προϊόντα, στις αγορές της Ευρώπης είναι πολύ μεγάλη, πράγμα το οποίο αποδεικνύει ότι δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε η ενιαία αγορά προς όφελος των καταναλωτών ή γενικά δεν διευκολύνει την αλυσίδα των προμηθειών και έτσι ίσως θα πρέπει να κοιτάξουμε, γιατί το συστήσαμε και σε ένα άτυπο γεύμα που είχαμε χθε. όπου ορισμένοι ε, λιανέμποροι πρότειναν μια ιδιαίτερη μνήα στις, στις διαφορές τιμών. Πρέπει να δούμε βεβαίως αν είναι ουσιαστικές, αν είναι σοβαρές διαφορές τιμών είναι κάτι το οποίο αφορά και τους συναδέλφους από την Ανατολική Ευρώπη, οι οποίοι επισημαίνουν ότι μπορεί από τη μια χώρα στην άλλη να υπάρχουν μικρές διαφορές μεταξύ των προϊόντων, χωρίς πάντα να υπάρχουν επιστημονικά ε, στοιχεία για το θέμα αυτό. Πολλοί από, όσοι, από όσους έχουν πάει σε αποστολή στις χώρες αυτές διαπιστώνουν κάποιες μικροδιαφορές στην ποιότητα. Άρα εκεί θα πρέπει να μιλήσουμε για ε, αγορά προϊόντων και όχι υπηρεσιών, αλλά ταυτόχρονα και για πιστοποίηση και για προδιαγραφές ποιότητας για τον καταναλωτή. Εδώ ίσως επεκτείνουμε κάπως το πεδίο των αρμοδιοτήτων μας. Εγώ πάντως θα καταθέσω τις σχετικές τροπολογίες. Επίσης για πρώτη φορά, αν δεν απατώμε, κατατίθεται μια τροπολογία για θέματα ε, του franchising που είναι ένας ε, σημαντικός τρόπος για ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και το οποίο franchising όταν λειτουργεί καλά μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην οικονομική δραστηριότητα. Ξέρετε ότι υπάρχουν πτυχές και ανταγωνισμού βεβαίως ε, και συμφωνιών μέσα από τις συμβάσεις αυτές που θα πρέπει να εξετάσουν πιο προσεκτικά, όρων δηλαδή στις συμφωνίες. Αλλά πάντως είμαι γνώμων που το θίγεται και πιστεύω ότι και οι συνάδελφοι θα ενδιαφέρονται να το δουν. Πρότεινω λοιπόν αυτές τις ιδέες για να προχωρήσουμε και για το ηλεκτρονικό εμπόριο η γενική προσέγγιση θα πρέπει να είναι η ενίσχυση της ανάπτυξης ενός ανταγωνιστικού τομέα που θα ενθαρρύνει και την είσοδο στην αγορά εργασίας και νέων ανθρώπων. Πάντως από την επίσκεψη στην Ελλάδα την προηγούμενη εβδομάδα είδαμε από τα στοιχεία των συνδικαλιστικών σωματείων και θα δημοσιευθούν αυτήν την εβδομάδα νομίζω ότι είναι πολύ ε, περιορισμένος ο ανταγωνισμός σε πολλούς τομείς της, ευρωπαϊκής, της ελληνικής αγοράς. Ε, εκεί που ιστορικά υπάρχουν φραγμοί στην είσοδο κάποιου σε έναν τομέα και ο κύριος Χαζηδάκης από ό,τι φαίνεται ο Υπουργός Ανάπτυξης σκοπεύει να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα. Τα έχει εξετάσει και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα από πλευρά τη και αυτά νομίζω σχετίζονται και με τα όσα είπα ω προ την ορθή λειτουργία τη αγορά. Άρα, όταν υπάρχει έλλειψη ανταγωνισμού για λόγου, σε παραδείγματι, γεωγραφικών ιδιαιτεροτήτων ή δραστηριότητε οι οποίε μπορεί να έχουν χαρακτηριστικά που αποθαρρύνουν κάποιον ε, νέο να, εισαχθεί στην αγορά, θα πρέπει ίσω να δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή. Ίσως θα μπορούσε η κυρία Κοράτσα να ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Ναι, και μια σχετικό με την έκθεσή της. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα. Τρεις συνάδελφοι ζητούν το λόγο. Σας παρακαλώ να είστε σύντομοι. Γιατί και άλλη συζήτηση θα δοθεί ευκαιρία να έχουμε και τροπολογίες μπορείτε να καταθέσετε. Κυρία Στάιλερ, Μπέλα, Πάντσερη. Έχετε το λόγο. Κυρία Στάιλερ. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και τον εισηγητή μας. Είναι πρόσδεκτη η προσέγγιση που παρουσιάσατε. Ναι, καθένα θέλουμε να στηρίζουμε ε, τέτοιες πρωτοβουλίες και ξέρω ότι στηρίξατε αυτή την εθελοντική πρωτοβουλία για τις καινοτόμες επιχειρήσεις. Υπάρχουν όμως και άλλα λεφτά συστήματα. Με την Επιτροπή, παραδείγματο χάρη αναφερθήκαμε στο τεστ ε, όπου ε, νεαροί επιχειρηματίες ε, συναγωνίζονται και χρηματοδοτούνται για να ιδρύουν την επιχείρησή τους. Έχουμε τα καταστήματα pop-up. Υπάρχουν τόσο πολλά διαφορετικά συστήματα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να έχουμε Φερρυπίν έναν ευρωπαϊκό ανταγωνισμό, δηλαδή ε, στο λιανικό εμπόριο βλέπουμε ένα πολύ μεγάλο πλούτο που διαθέτουν οι επιχειρηματίες και μπορούμε να ανταλλάσσουμε εμπειρίες. Ε, ξέρω ότι έχουν ένα, μια ομάδα υψηλού επίπεδου για το λιανικό εμπόριο που θα αρχίσει να συνεδριάζει το Δεκέμβρη. Καλό θα ήταν να ακούσουμε και τα σχόλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αυτήν την ομάδα. Επίσης, ε, το θέμα του ανεξάρτητου διαμεσολαβητή για τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές στην αλυσίδα τροφίμων. Ε, το ανέφεραν κάποιοι συνάδελφοι και ήθελα και εγώ να το σχολιάσω. Για την ομάδα δράση για το λιανικό εμπόριο θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μα ενημερώσει για το προς τα που κατευθυνόμαστε ουσιαστικά για τα πεπραγμένα. Ευχαριστώ και πάλι προς τον εισηγητή και θα τον βοηθήσουμε για να ευοδοθούν οι προσπάθειές του. Σας ευχαριστούμε κυρία Αμπέλα. Ευχαριστώ. Σε κάθε παρέμβαση που ακούσαμε, ακούστηκε ο όρος ηλεκτρονικό εμπόριο. Το σχέδιο δράσης για το λιανικό εμπόριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει πολλά θετικά στοιχεία, αλλά λείπει κάτι. Και θα μιλήσω και στα αγγλικά μιλώντας για τους μεγάλους λιανεμπόρους. Η μεγαλύτερη λιανέμπορη λοιπόν Πώς προσεγγίζει το θέμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι υπάρχουν ε, ουσιαστικά εμπόδια για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Αλλά τι γίνεται. Οι ίδιοι οι εμπορευόμενοι δεν μπορούν να επιλέξουν που θα διαθέσουν τα προϊόντα τους. Αυτό είναι αντίστοιχο προς αρχές της ενιαίας αγοράς. Αφήστε που συνιστά διακριτική μεταχείριση για τις απομακρυσμένες περιοχές όπως η Μάλτα. Κάποιοι αποκλείονται. Είδαμε και στην ακρόαση του Αρμοδίου Επιτρόπου ότι Υπάρχει πρόθεση να αναλυφθεί δράση για το θέμα των ε, μεγάλων λιανεμπόρων. Ελπίζω να μπορέσουμε να ασχοληθούμε και με αυτό. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ για αυτή τη γεωγραφική διακριτική μεταχείριση. Είναι ένα ζήτημα που συζητήσαμε στην ομάδα εργασίας ε, για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Είχαμε και στοιχεία από τα ε, ευρωπαϊκά και κέντρα καταναλωτών και έχουμε και διαθέσιμες πληροφορίες στον ιστότοπο, αν θέλετε να δείτε. Ο κύριο Παντσέρη τώρα. Ναι, ναι, ένα λεπτάκι θα μιλήσω μόνο, Πρόεδρε. Μετά από όλα αυτά που άκουσα, ε, μπορώ να πω ότι ε, ο κύριος De Jong εργάστηκε με εξαιρετικό τρόπο και συμφωνώ με την ε, πλειοψηφία όσων ακούσαμε μέχρι στιγμής. Δεν μπορούμε να ασχολούμαστε μόνο με τα οικονομικά ζητήματα και τις επανισορρόπησης της διανομής και το λιανικό εμπόριο ή ακόμη και μόνο με την απασχόληση. Επιτρέψτε μου κύριε Σιγητά να κάνω κι εγώ κάποιες προτάσεις για να έχουμε μια γενικότερη προσέγγιση. Υπάρχει μια σημαντικότατη κοινωνική πτυχή, διότι Λόγω των δημογραφικών εξελίξεων και της γύρανσης του πληθυσμού χρειαζόμαστε ε, τα, ε, το εμπόριο εγκύτητας, κυρίως από μακρισμένες ε, γειτονιές. Τώρα τι γίνεται στις μεγάλες πόλεις. το λιανικό εμπόριο αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα, αλλά είναι ένα απαραίτητο κοινωνικό στοιχείο και βασικός παράγοντας ανάπτυξης για πολλές πόλεις. Καλό θα ήταν ε, μέσα στην έκθεση μας να απευθύνουμε έκκληση προς ε, τις τοπικές αρχές, ούτως ώστε να υιοθετήσουν ε, ένα σχέδιο δράση ευνοϊκό για το λιανικό εμπόριο. Δεν θα παραβιαστούν οι κανόνες ανταγωνισμού, απλώ θα στηρίξουν το λιανικό εμπόριο που είναι απαραίτητο για την ευρωπαϊκή οικονομία. Ευχαριστώ. Έχει έρθει η κυρία Ρίζ Μέντα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν, δεν μπορώ κυρία Ρίμπε να σας δώσω πολύ χρόνο αλλά καλό θα ήταν να ακούσουμε κάποια γενικά σχόλια. Τι πιστεύετε για αυτή την έκθεση και ούτως ή άλλως θα έχουμε και πάλι μελλοντικά την ε, ε, ευκαιρία να συνεχίσουμε το διάλογο μας. Κάποιες καταληκτικές παρατηρήσεις αν θέλετε να κάνετε. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη λοιπόν. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω φυσικά τον εισηγητή για την εξαιρετική του έκθεση, η οποία ευθυγραμμίζεται σε μεγάλο βαθμό με τις σκέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για το σημαντικό αυτό τομέα που γνωρίζουμε ότι είναι πολύ σημαντικός και για την οικονομία αλλά και για την απασχόληση. Θα προσθέσω δε εγώ και για τις μικρές επιχειρήσεις. Πράγματι, στον τομέα του λιανικού εμπορίου υπάρχουν πάρα πολύ μικρές, πολύ μικρού μεγέθους επιχειρήσεις. Άρα το σχέδιο δράσης για το λιανικό εμπόριο απευθύνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Θα σχολιάσω μόνο ορισμένα από όσα συζητήσατε στις παρεμβάσεις σας και μετά θα μιλήσω για την ομάδα υψηλού επίπεδου. Για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Από ό,τι άκουσα, στο τέλος τουλάχιστον δεν βλέπω να υπάρχει τόσο μεγάλη διαφωνία ως προς ε, το ότι αναπτύσσεται αυτός ο κλάδος και γι' αυτό θα πρέπει να προσαρμοστούμε και υπάρχει ανάγκη στο σχέδιο δράσης ε, εξετάζουμε μεταξύ άλλων την καινοτομία, με επιχειρησιακά μοντέλα. Υπάρχει η πλατφόρμα για την καινοτομία και η Κομισιόν λαμβάνει υπόψη ε, τις ανάγκες των ε, πολύ μικρών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Όπως γνωρίζετε, είχαμε καταρτήσει ένα ξεχωριστό σχέδιο δράσης για το ηλεκτρονικό εμπόριο και εκπονήθηκε μια έκθεση υλοποίησης. Θα επανέλθω και στον μήνα νέας αγοράς. Μία από τις εβδομάδες του μήνα αυτού αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο. Είστε λοιπόν ευπρόσδεκτοι να συμμετάσχετε στις συζητήσεις ε, για την ενιαία αγορά και για αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Πολλές φορές ε, έγινε λόγος... Μισό λεπτάκι να βρω εδώ τις σημειώσεις μου. Α, ναι, μάλιστα. Για τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές. Θα ήθελα να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει την εθελοντική πρωτοβουλία των εμπλεκομένων φορέων. Είχαμε και εμεί συμμετάσχει στην ανάδυση, αν μπορώ να το πω έτσι, αυτής της πρωτοβουλίας και θα συνεχίσουμε να την υποστηρίζουμε. Αυτό είναι σαφές. Έχει γίνει σημαντική δουλειά τεράστιου μεγέθου από ε, τους ε, διαφερομένους φορείς που δεν θα πρέπει να υποτιμηθεί πόση προσπάθεια κατέβαλαν και επένδυσαν για να λειτουργήσει αυτή η θελοντική πρωτοβουλία και την χάνει τη περίπτωσης υποστήριξή μα. Από την άλλη πλευρά, διεξαγάγαμε διαβουλεύσεις ε, για την πράσινη βίβλο σε ό,τι αφορά το, τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές. Από εκεί ξεκάθαρα προκύπτει αυτό που είπε και ο κύριο Ντεγιό. Επιβολή. Επιβολή και εφαρμογή της νομοθεσίας. Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Υπάρχει πρόβλημα. Το εξετάζουμε πολύ προσεκτικά. Αυτή τη στιγμή εκπονούμε μια μελέτη αντικτύπου για την πράσινη βίβλο και μελετούμε τη, τα αποτελέσματα της διαβούλευσης και όλων, όλα τα άλλα έγγραφα που έχουμε λάβει και θα διατυπώσουμε τα τελικά μας συμπεράσματα για να δούμε κατά πόσον χρήζει μιας ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας η κατάσταση στο με αυτό. Δεν θα σχολιάσω διαμακρόν, αλλά θα έρθω σε μια μικρή λεπτομέρεια ή μάλλον όχι τόσο εδώ αλλά τέλος πάντων το cost selling είναι μια πάρα πολύ πολύπλοκη έννοια. Πολλές χώρες έμαθαν ότι προσπαθώντας να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα αυτά μέσω της νομοθεσίας μπορεί να ε, οδηγήσουν στη δημιουργία νέων ειδών στρέβλωσης και στις συστάσεις αναχώρα προς τη Γαλλία σημειώνει η Κομισιόν σε ό,τι αφορά την πόλη της πολύ σε χαμηλό κόστος, λόγω selling, ότι ναι μεν υπάρχει αυτός ο στόχος ε, να ε, υπάρχει στήριξη των παραγωγών και των μικρών αλυσίδων, αλλά θα μπορούσε αυτός ο στόχος να επιτευχθεί με λιγότερο παρεμβατικές ή στρεβλωτικές μεθόδους. Και πρέπει λοιπόν να το δούμε, να το δούμε πιο προσεκτικά. Η δικαιόχρηση, το franchising αναφέρθηκε πολλές φορές ε, από τη συζήτηση προέκυψε ότι υπάρχει ανάγκη να διευκρινιστεί έτσι περαιτέρω το ζήτημα αυτό. Και δεν είναι πάντοτε ξεκάθαρο περί τίνος πρόκειται. Αυτό θα πρέπει να το διευκρινίσουμε. και σε ό,τι αφορά τους ε, χωρικούς ε, περιορισμούς προμήθειας. Υπάρχει ένα πρόβλημα διαφορετικών τιμών που εφαρμόζεται. Διαφορετικές τιμές ε, από τους προμηθευτές στις διαφορετικές χώρες. Εμείς το εξετάσαμε με την Πράσινη Βίβλο και το εξετάζουμε και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο Αρμόδιος Επιτρόπος ε, δίνει προτεραιότητα στο θέμα αυτό. Δεν είναι εύκολο το θέμα αυτό. Είναι άκρος πολύπλοκο θα έλεγα μάλιστα. Δεν μπορούμε να τα βλέπουμε άσπρα ή μαύρα τα πράγματα. Κύριε Πρόεδρε, θα ολοκληρώσω εδώ λέγοντα ότι σε ό,τι αφορά την ομάδα υψηλού επίπεδου για, για το ελληνικό εμπόριο, είναι κάτι σημαντικό. Δείχνει ότι το σχέδιο δράση ε, δεν έγινε άπαξ κάτι το οποίο υλοποιήθηκε μία φορά και μετά έπαψε. Ε, δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε τη σημασία του λιανικού εμπορίου. Στόχος λοιπόν αυτής της ομάδας ψηλοεπέδου να παρακολουθεί την πρόοδο σε σχέση με αυτό το σχέδιο δράσης, αλλά και πέρα από αυτό να δει και τι μελλοντικές προκλήσεις υπάρχουν. Με βέβαια ότι θα λάβει υπόψη και τα δικά σας σχόλια για την κρίση, τις επιπτώσεις της κρίσης και τις μικροπιστές επιχειρήσεις. Σε ό,τι αφορά τη σύνθεση τη ομάδα, στο παρόν στάδιο δεν μπορώ να σα πω τίποτα, δεν έχει ακόμη συγκροτηθεί. Έχουμε όμω λάβει πάρα πολλέ ε, αιτήσει υποψηφιότητα από διαφορετικού ε, ενδιαφερομένου φορεί και ελπίζω να μπορέσουμε να σας πούμε περισσότερα σε σχέση με τη σύνθεση τη ομάδας αυτής ε, στο άμεσο μέλλον. Ευχαριστώ. Τα είπα λίγο συνοπτικά, λίγο περιληπτικά, αλλά δεν είχαμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μα. Πρώτα, σας ευχαριστώ πολύ. Λυπούμε, δεν είχαμε πολύ χρόνο πράγματι, το βιάσαμε λίγο το θέμα, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρετε όμως έχουμε σημαντικές ψηφοφορίες που έπονται. Ο Ντένις δεν θέλει να δευτερολογήσει, τον ευχαριστώ πολύ, έτσι εξοικονομούμε λίγο χρόνο παραπάνω. Να σας πω όμως εγώ τώρα το χρονοδιάγραμμα για να είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Προθεσμία κατάθεση τροπολέγων 10 Σεπτεμβρίου, την επόμενη εβδομάδα. Είχατε τη δυνατότητα να μελετήσετε την έκθεση από τον Ιούλιο, άρα δεν θέλαμε παραπάνω χρόνο. 25 με 26 Σεπτεμβρίου εξέταση τροπολογιών, 27 συμβιβαστική, 5 Νοεμβρίου ψηφοφορία και περιμένουμε και την έκθεση του Ντέιβιτ Κάζα από τη Μάλτα. Ίσως η κυρία Μπέλα θα μπορούσε να του πει ορισμένα πράγματα. 17 Οκτωβρίου είναι αυτή η έκθεση θα συνεισφέρει λοιπόν και η Επιτροπή Απασχόληση. Προχωρούμε. Ελπίζω να έχετε μαζί σα τις κάρτες ψηφοφορίας. Πρώτα απ' όλα, τι ψηφίζουμε, το Γενικό Προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το οικονομικό έτος 2014. Γκολ Πέλτς είναι η συγκητριά μας. Ε, δεν ξέρω, έχετε να κάνετε κάποια παρατήρηση πριν περάσουμε στην ψηφοφορία. Όχι, ωραία. Γραμματεία προτείνει να δω και αν συμφωνεί η Συγγήτρια ότι σε σχέση με αυτή τη λίστα ψηφοφορίας που έχετε, να ψηφίσουμε πρώτα τα κονδύλια του υπερπλογισμού, τις θέσεις του υπερπλογισμού. Άρα, σας παρακαλώ πρώτα να δείτε τη σελίδα 4, τα κονδύλια του προπολογισμού. Από τους σοσιαλιστές ποιος είναι συντονιστής. Α, η κυρία Στάιλ. Μπορούμε όλες μαζί, όλα μαζί τα κονδύλια να τα ψηφίσουμε. Ωραία. Όλα μαζί λοιπόν στην τέταρτη σελίδα ψήφι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται με σαφή πλειοψηφία. Σας ευχαριστώ και τώρα περνάμε στο ψήφισμα. Ξεκινάμε με την τροπολογία 1, κάμεν, ψήφι υπέρ. Κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 2 Σμιτ υπέρ, κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ, κατά απορρίπτεται. Τροπολογία 4 υπέρ, κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ, κατά απορρίπτεται. Τροπολογία 6 υπέρ, κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 7, για να δούμε. Καταπίπτει. Όχι, δεν καταπίπτει. Ψηφίζουμε την 7, είναι συμβατή με την 6. Νομίζω. Λοιπόν, ψήφι υπέρ τη 7. Κατά. Να ελέγξουμε καλύτερα, δεν είμαι βέβαιος, γιατί δεν έχω δει αν είναι όλοι εδώ. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 7 Σμιτ. 28 είναι η ε, Ωραία, 15 υπέρ, 12 κατά εγκρίνεται σαφώς. Τροπολογία 8 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 9 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 10 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 11 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 12 αποσύρεται. Τροπολογία 13 υπέρ, κατά, Απορρίπτεται. Όχι. Εγκρίνεται. Θέλετε να το ελέγξουμε. Ας ελέγξουμε λοιπόν την τροπολογία 13. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. 16 υπέρ, 13 κατά, 29 ψηφίσαντε. Αυτή τη φορά τροπολογία 14 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 15 υπέρ, κατά, αποχέ, ε, εγκρίνεται. 16 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 17 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 18 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 19 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Και τώρα ηλεκτρονικά ψηφίζουμε το σύνολο της ΕΚ της γνωμοδότησης. Άρχεται η ψηφοφορία. 29 βουλευτές ψηφίζουν. Πέρας ψηφοφορίας 25 υπέρ 2 κατά μια αποχή. Σας ευχαριστούμε κύριε Γκάλ Πέλτς. Και ελπίζουμε να προσπίσετε την θέση μας των υπολογισμών. Ευχαριστούμε και περνάμε, ναι, να σας πω ποια ε, θέματα ακολουθούν. Τρεις σημαντικές εκθέσεις στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων. Τα παρακολουθείτε τα θέματα αυτά, φαντάζομαι, του σύνεγγυς. Είχαμε εκθέσεις αναφορές για την εξέλιξη ε, των πραγμάτων τουλάχιστον δύο-τρεις φορές, έχουμε κάποιες αλλαγές, αλλά συνολικά μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι και με τις τρεις εκθέσεις, επειδή είναι σημαντικό το θέμα, θα δώσω το λόγο στους εισηγητές και στους σκιώδεις που θελήσουν τον λόγο ενδεχομένω. Αλλά στους εισηγητές πρώτα απ' όλα. Μάρκ Ταραμπελά, ο πρώτος, γιατί έχουμε δύο ψηφοφορίες. Έχεις τον λόγο. Merci, Président. En effet, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα είναι σύντομη η ψηφοφορία το Δεκέμβρη και τον Ιανουάριο. Μας πήρε πολύ χρόνο, αλλά καταφέραμε να καταλήξουμε τότε σε συμβαστικέ τροπολογίε για τις τρεις εκθέσεις, για τις δύο δικέ μου και τη μία του κ. Ζουδά. Ε, δεν χρειάζεται να μακρηγορήσω για το περιεχόμενο. Στην Ολομέλεια ενδεχομένω να επανέλθω με κάποιε λεπτομέρειε. Ε, ίσως ε, ζητήσω από κάποιον από την ομάδα μου, αλλά για το περιεχόμενο ίσως επανέλθω για τα, ε, τις κοινωνικές συμβάσεις ε, για την εξωτερική ανάθεση και την υπεργολαβία την πλέον συμφέρουσα προσφορά ε, τις τιμές που είναι με μη φυσιολογικό τρόπο χαμηλές οι πρακτικές της αναθέτουσας αρχής των εμπορικών φορέων σε όλα αυτά έχουμε σημειώσει πρόοδοι, κοινωνικές υπηρεσίες, θα μιλήσω και για αυτές, ε, διότι θυμάστε το αμφιλεγόμενο άρθρο 17.2 που πλέον δεν υπάρχει καταργήθηκε, αλλά θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί γιατί θα επιπτύσει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών να μεταγράψουν σωστά στην εθνική τους νομοθεσία τις διατάξεις και να έχουν ευελικτέ δημόσιες υπηρεσίες για την ανάθεση. Ήθελα μόνο να σας πω, Πρόεδρε, ότι ακόμη μια φορά θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, για όλη αυτή τη δουλειά τους και όσες ηγητές. Ενάμιση χρόνο εργαστήκαμε. Ο κύριος Έγγελ, ο κύριος Κρόιτσμαν, η κυρία Ρουλέ που συνέδεσε συνέταξε την έκθεση πρωτοβουλία, ο κύριος Ντε ε, δεν πρέπει να ξεχάσω κανέναν. Όχι, ξέχασα τον πρόεδρο. Δεν σας, δεν σας ξέχασα ουσιαστικά, ε, γιατί με, είστε πρόεδρος της Επιτροπής ΙΜΚΟ, φυσικά πέρα από την ιδιότητα του εισηγητή και ήθελα να σας συγχαρώ και σας, διότι ίσως αυτό είναι άσχημο, ναι, ότι μετά τη θητεία θα βγείτε στη σύνταξη. Αυτή είναι η πρόθεσή σας. Ε, και πραγματικά με πάσα ειλικρίνεια σας ευχαριστώ για τον τρόπο που καθοδηγήσατε τη συζήτηση στο Συμβούλιο. Δεν συμφωνούσαμε όλοι για τις διάφορες έννοιες, για τους ορισμούς και χαιρετώ και εσάς και τους κοιόδους εισηγητές διότι ε, πριν από κάθε συνάντηση, πριν από κάθε σύσκεψη των σκιωδών προετοιμαζόσασταν με τόσο αποτελεσματικό τρόπο. Θα μπορούσα να μιλήσω για τον Τόνιο Πανσέρη και τον ε, Φιλίπ Σουμβάν γιατί κάναμε και κοινέ ε, συνεδριάσεις. Ε, υπήρχε μεγάλη συνέπεια στο Κοινοβούλιο φυσικά στι διαπραγματεύσει ε, κέρδισε ε, σε πολλά σημεία το Συμβούλιο, αλλά πάντως ε, μιλούσε με μία φωνή το Κοινοβούλιο και επίση ήταν εξαιρετική η προετοιμασία που κάναμε πριν από τι συσκέψει. Επίση, να ευχαριστήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που, α μην το ξεχνάμε, στι 21 Δεκεμβρίου 2011 κατέθεσε την αρχική πρόταση. Ήταν ούτως ή άλλω καλή η αλλω καλη η πρόταση, την επιβεβαιώσαμε για κάποια επιμέρου σημεία γιατί ήταν σημαντικό να είναι είναι ηχηρό το μήνυμά μας και ας μην ξεχνάμε ότι η έκθεση αυτή είναι σημαντική διότι μιλάμε για το 19% του ΑΕΠ της Ευρώπης. Χρειαζόταν λοιπόν για την αναθεώρηση της οδηγίας να μεριμνήσουμε ώστε να επενδύονται καλύτερα τα δημόσια κονδύλια και πιστεύω ότι τα καταφέραμε. Εργαστήκαμε ε, με αποθελισματικό τρόπο. Δεν γεννήθηκε το 8ο θαύμα του κόσμου, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ξεκάθαρο το μήνυμα που περνάμε και στις δημόσιες αρχές αλλά και στους εμπορικούς φορείς που ανταγωνίζονται για τις κρατικές προμήθειες και ε, να ευχαριστήσω και το προσωπικό τους βοηθούς μας, ε, ε, τη Μαρή Μπουό που ξεκίνησε και την Αλέσια Νταμπό που ακολούθησε μέχρι τέλους το φάκελο και κυρίως κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Φυσικά να πω καλά πράγματα για τη Σαντίνα Μπατολέτσι από την δική μου πολιτική ομάδα. Ήταν πολύ δύσκολες οι διαπραγματεύσεις. Ε, να ευχαριστήσω και το επιτελείο του ε, Κοινοβουλίου. Ήταν δυσχερέστατο το έργο μας, δεν έχουμε τέτοια στελέχωση όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο. Παρ' όλα αυτά τα καταφέραμε και είναι ξεκάθαρο το μήνυμα. Μακρηγόρησα παρόλα αυτά νομίζω, αλλά αξίζει γιατί κάναμε ε, δεκάδες συνεδριάσεις, εκατοντάδες ώρες, τόνους χαρτιού, δεν πρέπει να το λέμε βέβαια αυτό, και 1,5 χρόνο εργασιών, οπότε είναι φυσιολογικός. Ευχαριστώ όλες και όλους για την την αγαστή συνεργασία. Ε, σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ήταν μεγάλη χαρά. Θα είναι μεγάλη η πρόκληση, φαντάζομαι, ίσως όχι τόσο μεγάλη όσο τα, οι δημόσιες συμβάσεις πέραν των παραχωρήσεων που ήταν οπωσδήποτε πολύ φιλόδοξη. Ας ακούσουμε λοιπόν τον συνάδελφο. αλλά επισημαίνω ότι τις παραχωρήσαμε μια δομή πολύ ογκώδη. Ας ακούσουμε λοιπόν τον συνάδελφο να μας πείτε δύο λόγια για τη δική σας έκθεση. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να παρηγορήσω τον, τον συνάδελφο εισηγητή μόνο. Δεν είναι υπαρκτά πλέον τα θαύματα του κόσμου, τουλάχιστον όχι όλα. Γι' αυτό μην επιδιώξεις και εσύ να φτιάξεις άλλο ένα. Τι κάναμε ως προς την οδηγία αυτή. Φτιάχνουμε ένα ευρωπαϊκό νομοθέτημα για τις ε, παραχωρήσεις ε, σε θέματα έργων. Είχαμε βέβαια την οδηγία για τα μεγάλα έργα και τις βασικές αρχές συνθήκες συνθήκες, ιδιαίτερες συνθήκες και νομίζω ότι έτσι μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι γιατί βλέπουμε ότι τίθεται ένα τέρμα πλέον σε μια σειρά από ε, κειμενόμενα νομολογιακά συμπεράσματα και μπορούμε να έχουμε μια βάση πιο στερεή και εμείς βέβαια αλλά και οι επιχειρήσεις και πρέπει να πούμε ότι πολύ συχνά χρειαζόταν να περιμένουμε την ερμηνεία του δικαίου να τη δώσει ένας δικαστής. Άρα λοιπόν πλέον αποφασίζουμε, θεσπίζουμε δίκαιο, κάνουμε μια πρώτη πρόταση για ένα νομικό καθεστώς, χωρίς να θέλω να υψέλθω σε κάθε λεπτομέρεια και σε κάθε άρθρο ήταν ε, μακρά η περίοδος των διαβουλεύσεων, οι εργασίες, τα έγγραφα. Φτάνουμε πάντως σε ένα κείμενο με καλή, ε, καλές ισορροπίες. Υπενθυμίζω ότι είχαμε μεγάλη απόσταση στις θέσεις μεταξύ μας, αυτό το σημείο αφιτηρίας, και καταλήξαμε σε μια πολιτική θέση, γενική συμφωνία, η οποία θα επιτρέψει, πιστεύω, την ε, αποδοχή του κειμένου από τους πάντες. Θα πρέπει να θεωρηθεί δηλαδή ικανοποιητικό. Δεν ήταν τέλειο, αλλά πάντως έγινε πολύ καλή δουλειά και ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που συνεργάστηκαν, τους και ηγητές, που βεβαίως θέλω ρητά να αναφέρω, το Σνάλφο Χάρμπορ, τον συνάδελφο Παντσέρι, τη Ζόιλ, Ορλό, Χέντελ. Επίσης ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ομάδα του Μισελ Μπαρνιέ που δραστηριοποιήθηκε ιδιαίτερα στο θέμα αυτό και επίσης το προσωπικό μας και εγώ το δικό μου ε, προσωπικό ιδιαίτερα την Καρίν Μονφόχ βοηθό μου αλλά και την τεχνική ομάδα του ΕΚ που με βοήθησαν πολύ. Κάναμε πολύ δουλειά λοιπόν κύριε Πρόεδρε χρήσιμη πιστεύω. Και εάν ε, δεν φτάσαμε στο έπακρο των απαιτήσεών μας, πάντως μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι διότι θέσαμε ένα πρώτο λιθάρι στο δρόμο αυτόν και μπορούμε να προχωρήσουμε κοιτώντα με αισιοδοξία προς το μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, ο Πρόεδρος. Και εγώ καλωσορίζω εδώ τον, την εκπρόσωπο της Επιτροπής. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Και συνεχίζουμε με την ψηφοφορία. Ηλεκτρονικά όπως είπαμε. Ψηφίζουμε. Ηλεκτρονικά παρακαλώ. Πέρας. 27 υπέρ, μία ψήφος κατά, μία αποχή. Εγκρίνεται. Το επόμενο θέμα. Με το ίδιο αποτέλεσμα και στις παραχωρήσεις. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 26 2 κατά μία αποχή. Σας ευχαριστώ όλους Και θα να ευχαριστώ τα μέλη της Επιτροπής μας που είναι εδώ. Βλέπετε την Αλεξάνδρα, τη Ζούλια. Καλώς ήρθατε. Και όλους όσοι ήταν βέβαια παρόντες και βοήθησαν στην υπόθεση αυτή. Ευχαριστούμε θερμά. δεν ξέρουμε πότε θα πάει στην Ολομέλεια το θέμα. Θα κοιτάξουμε το χέτερο δυνατό. Και θα σας ενημερώσουμε. Και τώρα προχωρώ στο επόμενο θέμα. Η κυρία Ρόιτοβα δεν είναι εδώ. Γιατί δεν ψηφίζουμε το νέο νομοθετικό πλαίσιο, είχατε πει. Είσαστε εδώ τώρα, κύριε Ρόιτοβα. Θέλετε να γράψετε το λόγο. Να σας ενημερώσω όμως πρώτα γιατί δεν ψηφίστηκε. Όχι. Η κυρία Ρόιτοβα. Πρόεδρε, βλέπω μια σειρά από αναβολές. Και πρόκειται για μια οδηγία η οποία έχει μεγάλη σημασία. Πρέπει να προσδιοριστούν οι κανόνες της. Δεν θεωρώ ότι είναι σωστό να αναβάλλεται διαρκώς. Και έτσι θεωρώ ότι η Άννα δεν μπορεί σύντομα να λάβει μια απόφαση το Συμβούλιο, καλό θα είναι να αποφασίσουμε εμείς και με βάση τόσο που αποφασίσουμε να κάνουμε τη συνάντηση με την Προεδρία. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος. Ναι, υπάρχουν κάποια αναθεωρημένα κείμενα που μας έχουν ε, κατατεθεί ως βάση διαπραγμάτευση, αλλά από την άλλη αντέδρασαν ε, κάποια από τα κράτη-μέλη και αν έτρεψαν αυτή τη ισορροπία, προσπαθούμε να έρθουμε σε επαφή με την Προεδρία για το δούμε. Πάντως δεν είναι ικανοποιητική κατάσταση. Και πάμε στο επόμενο θέμα για ψηφοφορία. παρακαλώ την Επιτροπή να εγκρίνει μια προφορική ερώτηση που έχουμε συμφωνήσει με τους συντονιστές. Ευρωπαϊκή αγορά και Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος, Ελβετία. Το κείμενο το έχουν συζητήσει και διαπραγματευτεί οι πολιτικές ομάδες. Δεν ξέρω αν ο κύριος Φαπ θέλει το λόγο. Μπορούμε να εγκρίνουμε. Προφορική ερώτηση παρακαλώ υπέρ. Δεν χρειάζεται. θέλουμε να κάνουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία καλύτερα για το κείμενο της προφορικής ερώτησης. Και έτσι πάει στην, ε, στις υπηρεσίες Ολομέλειας για κατάθεση προφορική ερώτηση και περνώ στην γνώποδότηση του κυρίου Κοφεράτη για το 2020. Κάρση 2020 για να δούμε. Cars 2020, ισχυρή ανταγωνιστική βιώσιμη βιομηχανία. Α πάρουμε τι ε, κάρτε μα. Πρόκειται για έγκριση. Ψηφίζουμε απευθείας. Δεν είναι εδώ ο κ. Κοφεράτη λογια συμβαστική πρώτη υπέρ κατά εγκρίνεται. 3 και 4 καταπίπτουν. 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προφορική. Στην 8 του κ. Μπόρισοφ στον κατάλογο των ψηφοφοριών τον έχει ζητήσει ο εισηγητής την προφορική 8 λοιπόν υπέρ, κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ, κατά. Εγκρίνεται. 4 συμβαστική υπέρ, κατά. Εγκρίνεται. 5 υπέρ, κατά. Εγκρίνεται. 6 υπέρ, κατά. Εγκρίνεται. 19 υπέρ, κατά. Απερίφθη. 20 του εισηγητού υπέρ. Ας επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Α, συμφωνείτε μάλιστα. Καλώς. 20 λοιπόν. Κατά. Έγκριθηκε. Συμβαστική 7 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 25 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 8 υπέρ κατά εγκρίνεται 27 υπέρ κατά ε, 30 υπέρ κατά απερίφθη συμβαστική 9 σε τμήματα που ζητούν η δική μου ομάδα συντηρητικοί μεταρρυθμιστές Πρώτο κομμάτι, η συμβαστική τροπολογία εκτός των λέξεων συμπεριλαμβανομένης νομοθετικής πράξεως. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Και τώρα οι λέξεις αυτές, οι φράσεις συμπεριλαμβανομένης νομοθετικής πράξεως. Υπέρ, κατά. Απερίφθη. Δεν χρειάζεται να επαληθεύσουμε νομίζω. 35. Μπορισόφ. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 36 Βέστφαλ. Υπέρ. Κατά. Ας επαληθεύσουμε. Τροπολογία Βέστφαλ. Άρχεται. Πέρασε. Απερίφθη με μία ψήφο διαφορά. 14 υπέρ 15 κατά συμβαστική 10 υπέρ κατά εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ κατά εγκρίνεται. 42 υπέρ 42, έκανα λάθος λέω, πρέπει 42 υπέρ κατά εγκρίνεται συμβαστική 12 υπέρ κατά εγκρίνεται 45 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 46 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται 47 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται 48 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται 49 υπέρ. Κατά. Ας το κοιτάξουμε αυτό άλλη μια φορά. Τη 49 την επαληθεύουμε. Ψηφίσει κανεί άλλο. Ψήφισαν όλοι. Εγκρίνεται. 16 υπέρ, 12 κατά. 50 υπέρ, κατά. Εγκρίνεται. 51 υπέρ, κατά. 51 να υπερθέσουμε. Εγκρίνεται μία ψήφος διαφορά. 52 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Σε θεολογικές αναφορές, τροπολογία 1, κοφεράτη. Υπέρ. Κατά αποχές. Ας επαληθεύσουμε την υπαριθμόν 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Απερίφθη. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά εγκρίνεται το σχέδιο γνωμοδότησης παρακαλώ ηλεκτρονικά ψηφίστηκαν, ψήφισαν όλοι. 29 κάρτε έχω στο σύστημα, αλλά δεν βλέπω να έχετε ψηφίσει όλοι, τρέπεστε. Καλώ πέρε προφορίε. 26 υπέρ, μία ψήφο κατά, μία αποχή εγκρίνεται. Και τώρα πάμε στην έκθεση του κυρίου Σφάπ για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο για το στονισμό των, της οικονομικής πολιτικής. Θέλετε το λόγο. Θέλω μία ερώτηση να κάνω, διότι τώρα θα ψηφίσουμε αυτή τη γνωμοδότηση και πρέπει να έχουμε κατά νου ότι υπό την ηγεσία μου, αλλά χάρη στην ανακοίνωση του Επιτρόπου Μπαρνιέ, η Επιτροπή μας άρχισε να εμπλέκεται ε, ενεργά με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και θα ήθελα να μου το επιβεβαιώσετε αν ισχύει η σοφή διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε να διακόψει τις δραστηριότητες αυτής της δραστηριότητας της Επιτροπής μας σε σχέση με το Ευρωπαϊκό ε, Εξάμεινο. Εγώ πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ καλό για την ενιαία αγορά. Μπορείτε να μου το επιβεβαιώσετε, ισχύει αυτό, ευσταθεί. Πρόεδρος. Ε, δεν ε, με συμβουλεύτηκε η διάσκεψη των Προέδρων για αυτό το ζήτημα. Ποτέ δεν ε, συζητούν άμεσα ούτως ή άλλως με τους Πρόεδρους των Επιτροπών. Αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσω εξ αρχής. οπότε η διάσκεψη των Προέδρων αυτοδιαβουλεύεται, θα το πω έτσι, και εκπρόσωποι των δύο κυρίως μεγαλύτερων πολιτικών ομάδων στη διάσκεψη των Προέδρων ζήτησαν ε, είναι οι μόνοι που μπορούν ε, μάλλον να υποστηρίξουν το έργο μας. Θα πρέπει να το ζητήσετε από αυτούς ε, που ούτως ή άλλως επικρατούν εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πέρα από αυτά τα πασαλήματα που κάνουν οι φιλελεύθεροι από εδώ και από εκεί και δεν μιλάω για την ποιότητα των εργασιών τους, μιλάω για τα αποτελέσματα των προσπαθειών τους. Τέλος πάντων, καλό θα ήταν να πάτε να ε, κυκλοφορήσετε και να μιλήσετε με τους συντονιστές των δύο μεγαλύτερων πολιτικών ομάδων. Ε, αν οι συντονιστές μου αναθέσουν εντολή να το κάνω, και εγώ μπορώ να το επισημάνω στην διάσκεψη των Πρόεδρων την ε, λανθασμένη απόφαση τους, αλλά δεν μπορώ να εγγυηθώ τίποτα. Μπορεί να θεωρήσουν ε, ότι το παρακάνουμε, ε, παρότι εμείς ασχολούμαστε με την ενιαία αγορά, ότι δεν θα έπρεπε να είμαστε το, να μένουμε τόσο πολύ και να επεμβαίνουμε τόσο πολύ. Λοιπόν, θα με βοηθούσατε σε αυτή την ε, εκστρατεία μου αν είχα την πλειοψηφία. Ας ψηφίσουμε τροπολογία 1. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 1. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Κατά τμήματα. Κυρία Κομφεράτη, πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Θα πρέπει να κάνουμε μια επαλήθευση. Το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 4. Παρακαλώ. Πέρας. Απορρίπτεται. Ε, τροπολογία 5 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Η 7 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Η 8 υπέρ. Ηλεκτρονική παρακαλώ για την 8. Uh, ε, the vote is closed. Πέρας. Απορρίπτεται. Η 9. Υπάρχουν διάφορε γλωσσικέ εκδοχέ. Το είπα υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Συμβαστική 12 υπέρ, κατά, Εγκρίνεται επίση. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την γνωμοδότηση. Για την έκθεση, διορθώνει ο πρόεδρο. Όχι, είναι γνωμοδότηση. Τι είναι. Ψήφισμα. Πέρα. 25 ψήφοι υπέρ μία κατά και τρεις αποχές. Εγκρίνεται. Ε, περιμένω λοιπόν το αίτημά σα, το οποίο εγώ θα διαβάσω συνέχεια στη διάσκεψη των Πρόεδρων και θα τα πούμε στην επόμενη σύσκεψη των συντονιστών. Και ο κύριος Σμιτ μπορεί να χαιρετήσει τον ε, ηγέτη της ε, ομάδας του. Μην με παρανοηθούν αυτά που είπα εγώ για την ποιότητα, το, την αποτελεσματικότητα μάλλον των εργασιών ε, των φιλελευθέρων. I am listed λόγω του χρονοδιαγράμματος, αντί να ασχολούμαστε με το σύνολο της έκθεση. ασχολούμαστε μόνο με τις τροπολογίες. Κάνουμε λοιπόν μια κοινή προσπάθεια, όλες τι πολιτικές ομάδες μαζί. Θα ήθελα λοιπόν να τις ψηφίσουμε. Ας αρχίσουμε με τις παραγράφου. Η πρώτη, υπέρ. Κατά. Από, εγκρίνεται. Δύο. Υπέρ. Κατά. Ε, εγκρίνεται. Ε, ε, η τρία. Υπέρ. Τροπολογία δεν είναι παράγραφος. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται νομίζω, αλλά να το ελέγξουμε. Τρία πέρας. Απορρίπτεται γιατί είναι η 14 προς 14, τροπολογία 4 υπέρ. Ηλεκτρονικά παρακαλώ. Η τέσσερα. Πέρας. Εγκρίνεται 15 προς 13. Τροπολογία 5 υπέρ. Υπέρ. Το έλκτη είναι, υπέρ ή κατά. Κατά. Εσείς όμως είστε υπέρ. Α ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Για την 5. Για 5. Πέρας. Εγκρίθηκε. Η 6 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 7 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται 8 υπέρ. Κατά εγκρίνεται 9 υπέρ. Κατά εγκρίνεται 10 υπέρ. Κατά εγκρίνεται Μπορούμε όλες μαζί να τις ψηφίσουμε τις υπόλοιπες. Υπάρχουν αντιρρήσεις. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Υπέρ. Κατά. Εγκρίθηκαν όλες. Ε, τώρα θα τις καταθέσουμε στην Επιτροπή ΕΚΟΝ για να ενσωματωθούν στη δική τους ε, έκθεση. Γι' αυτό και δεν χρειάζεται να υιοθετήσουμε εμείς την έκθεση. Ο κύριος Σβάμπ δεν με ακούει. Κύριε Σβάμπ, είστε μέλος της ΕΚΟΛ. Και κύριε Σμιτ. Ούτε εκείνος με ακούει. Κύριε Σμιτ. Συνεργαστείτε σας παρακαλούμε με τον κύριο Σφάμπ για να ενσωματωθούν αυτές τις τροπολογίες που ψηφίσαμε στην τελική έκθεση. Ε, σχολείο του κυρίου Σμίτ εκτός μικροφώνου, μα μη με παραξηγείτε, είμαι υπέρ του αρχηγού των φιλελευθέρων. Λοιπόν, για πάμε τώρα στη, στο επόμενο θέμα. Θα ήθελα να σε ενημερώσω ότι εχθέ συναντήθηκα με την ε, κυρία Τράουτμαν που είναι η συγγήτρια στην Καθήλυνα Αρμόδια Επιτροπή και την κυρία Φερχέγεν που είναι η σκιώδης δεν είναι εδώ νομίζω αλλά συμφωνήσαμε για διάφορες συμβαστικές τροπολογίες και υπάρχει με κάτι που συμφωνήσαμε μετά τις συζητήσεις, κυρία Στράτου, να το διαβάσω γιατί δεν νομίζω να το έχετε στους φακέλους, για την τροπολογία 4, πιο συγκεκριμένα, οπότε να έχετε το νου σας. Ας προχωρήσουμε. Η κυρία Φεχίγεν ήταν η μόνη σκιώδης που υιοθέτησε δικές μου τροπολογίες για την έκθεση. Την ευχαριστώ. Τροπολογία 2. Υπέρ κατά. Εγκρίνεται. 3 υπέρ κατά. Εγκρίνεται. Θα σας διαβάσω τώρα την τροπολογία 4, προφορική τροπολογία. Ε, συμφωνήσαμε με την κυρία Φεχέγιν και ελπίζω να συμφωνήσετε κι εσείς. Ε, σχετίζεται με τα θέματα της ουδετερότητας του δικτύου ε, και η Επιτροπή Βιομηχανίας ασχολείται με αυτό το θέμα. Τονίζει λοιπόν ότι η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων για την ποιότητα των υπηρεσιών κατά τη διαστολή με τον τρόπο διανομής μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα ε, και καλεί την Επιτροπή και τις ρυθμιστικές αρχές να παρακολουθήσει την κατάσταση και αν χρειαστεί να παράσχουν τα εργαλεία του άρθρου 42 της Οδηγίας για τις καθολικές υπηρεσίες ε, και αν χρειαστεί να εξετάσουν εξετάσουν το ενδεχόμενο υιοθέτηση επιπροσθέτων νομοθετικών μέτρων. Το καταλάβατε όλοι, επαντηρήσει όχι, ωραία, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Η τροπολογία 5, αυτή η προφορική τροπολογία που σα διάβασα, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Ε, η 6 υπέρ, κατά, ε, με την προφορική τροπολογία που έχει εγκριθεί, τροπολογία 7 υπέρ κατά εγκρίνεται, τροπολογία 8 υπέρ κατά εγκρίνεται, τροπολογία 1 υπέρ κατά εγκρίνεται ε, και τώρα θα ψηφίσουμε για την ίδια την έκθεση, παρακαλώ ηλεκτρονικά. Ε, ψηφίζει κανένας άλλος. Όχι, αρέσει σε όλους. Πολύ ωραία. 25 ε, ψήφοι υπέρ, μία αποχή, καμία ψήφος κατά. Σας ευχαριστώ πολύ για την εμπιστοσύνη που μου δείχνετε και θα φροντίσω ώστε να ενσωματωθούν αυτά στην έκθεση Επιτροπής Ανταγωνισμού και ευχαριστώ την κυρία Φερχέγιν για την προφορική τροπολογία. Τέρμα, τελειώσαμε με τις ψηφοφορίε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα νέα ε, γνωμοδότηση ε, με αποδέχνει την Επιτροπή ε, Εξωτερικών Υποθέσεων η κυρία Γκάλ Πέλτσιν, η συγγήτριά μας, για την τεχνολογική και βιομηχανική βάση της Ευρωπαϊκής Άμυνας. κυρία Γκάλ μπορείτε να μας παρουσιάσετε την, το σχέδιο γνωμοδότησης. Η κυρία Στάιλερ, ποιος άλλος Ποιος ε, άλλος σκιώδης είναι εδώ. Η κυρία Γκέπχαρτ δεν είναι εδώ που είναι σκιώδης. Δεν έχουμε Α, δεν έχουν διοριστεί ε, ακόμη οι ε, Βάιλερ Σμιτ, εγώ μπορεί να το σχολιάσω. <laughs> Είστε υποσκιασμένοι, δεν έχετε αρκετές σκιώδεις. Παρουσιάστε το σχέδιο γνωμοδότησης. Έχουμε την κυρία Σίλβια Καντσιούμπα από την Επιτροπή. Καλά τα λέω. Ωραία. Θα σας ακούσουμε μετά. Και μετά θα ξανακούσουμε την κυρία Γκαλπέλτς. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε δεν υπάρχουν αρκετοί σκιώδεις ηγητές, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το θέμα δεν είναι σοβαρό. Ε, το αντίθετο, είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. από στρατηγικής ε, πολιτικής πλευράς έχουμε συνεχώς αλλαγές και θα πρέπει βέβαια να αναζητήσουμε απαντήσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε η τεχνολογική βάση και η βιομηχανική βάση της Ευρωπαϊκής Άμυνας να μπορέσει να προχωρήσει. Θα ήθελα να ξεκινήσω με κάποια συγκριτικά στοιχεία στην κοινή Κίνα, Ιαπωνία και Ρωσία μαζί. Οι δαπάνες, οι αμυντικές δαπάνες είναι ε, ίσες με το άθροισμα των αμυντικών δαπανών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχουν 400.000 ε, ε, θέσεις εργασίας που τίθεται σε κίνδυνο για να καταλάβετε πόσο ε, είναι το μέγεθος αυτού του τομέα. Μιλάμε για εκατο εκατομμύρια ε, τζίρο. Καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη είναι η σημασία του τομέα αυτού. Δεν έχω βέβαια ακόμη λάβει το έγγραφο της Κομισιόν, αλλά μπορώ να σας πω ότι φαίνεται να υπάρχουν αλληλεπικαλύψεις στα έγγραφα της Κομισιόν σε σχέση με το δικό μου ε, έγγραφο. Πάντω αφετηρεί είναι η ίδια στους προπολογισμού των κρατών μελών. Το μερίδιο των αμυντικών δαπανών μειώνεται σταθερά. Ωστόσο, θα πρέπει η ανταγωνιστικότητα να βελτιωθεί. Ακριβώς για αυτό το λόγο η ανταγωνιστικότητα λοιπόν της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Μηχανίας πρέπει να βελτιωθεί και αυτό απαιτεί μεγαλύτερη και στενότερη συνεργασία και πιο ανοιχτό πνεύμα, μεγαλύτερη διαφάνεια στην αγορά, την αμυντική. Τις παρατηρήσεις μου τις εστιάζω σε έξι σημεία και θα σας δώσω σύντομα κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες πάνω σε αυτά τα σημεία. Πρώτα απ' όλα, ήδη συζήτησαμε τους κανόνες των δημοσίων προμηθειών και το πόσο διαφορετική είναι από τη μια χώρα στην άλλη. Αυτό παρεμποδίζει τη βελτίωση των επιδόσεων του τομέα. Βέβαια, σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να μιλήσουμε για ενιαία ε, αμυντική αγορά στην Ευρώπη. Υπάρχει μεγάλος κατακαιρματισμός, ε, υπάρχουν επικαλύψεις, παράλληλες διαδικασίες και όλα αυτά πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Επίσης, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να προωθήσουμε νέε τεχνικέ καινοτόμε τεχνικές στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων. Εξορθολογισμό. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τελευταίες εξελίξεις, στην ε, τεχνολογία εχμής. Θα πρέπει επίσης να προωθήσουμε και να δώσουμε κίνητρα για, μεγαλύτερη, για περισσότερη έρευνα και ανάπτυξη. Υπάρχει κάτι ακόμη που πρέπει να συζητήσουμε και το οποίο επηρεάζει τα μάλλον την αμυντική βιομηχανία. Είναι οι συμβάσεις, ε, τα τέφη δημοπράτησης, όλα τα σχετικά με τους διαγωνισμούς έγγραφα. Είναι τόσο πολύπλοκα και στη διατύπωσή τους που καθιστούν πάρα πολύ δύσκολους ε, τους διαγωνισμούς. Θα πρέπει κάτι να κάνουμε υπάρχουν δυσανάλογες τεχνικές απαιτήσεις ε, και εμπόδια τα οποία πρέπει να αρθούν ή τουλάχιστον να ελαχιστοποιηθούν. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι, είναι ιδιαίτερα αγαπητές αν θέλετε, ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα, αλλά ο τομέας αυτό ο αμυντικό, επειδή υπάρχει αυτή η ε, διάσπαση ο τη χώρας, δεν είναι ακριβώς φιλικός προς τις μικροπεσαίες επιχειρήσεις, υπάρχει έλλειψη ε, πρόσβασης στο κεφα... σε κεφάλαια και αυτό δυσκολεύει τα πράγματα στις... Ε, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν μπορούν εύκολα να έχουν πρόσβαση στην αμυντική αγορά. Θα μπορούσε να γίνει εδώ μια προσπάθεια να δημιουργηθεί μια εταιρική σχέση, όπως έχει γίνει σε άλλους τομείς. Ίσως θα μπορούσε η Κομισιόν να διευκολύνει την πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Αμυντική Βιομηχανία με μια πρόταση που θα υποβάλει προς αυτήν την κατεύθυνση. Επίσης, θα ήθελα να στήσω από την Κομισιόν και τα κράτη-μέλη να συνεργάζονται μεταξύ τους και με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας ε, για να προωθήσουν την ενσωμάτωση στον ευρωπαϊκό αμυντικό τομέα και των μικρότερων κρατών σε αυτή την ε, βιομηχανική τεχνολογική βάση της Ευρωπαϊκής Άμυνας για να ανοίξουν νέοι ορίζοντες για συνέργειες. Αυτή είναι οι συστάσεις που είχα να κάνω, πάρα πολύ συνοπτικά. Φυσικά και αναμένω τα σχόλια της παρατηρήσης σας, τις τροπολογίες είτε από τους Σκιώδης είτε και από οποιοδήποτε άλλο παρόντα σήμερα εδώ συνάδελφα. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ για να δούμε ποιος θα θέλει τώρα να συμμετάσχει στη συζήτηση. Βλέπω την κυρία Βάιλερ, βλέπω την κυρία Ρούλε, τον κύριο Σβά, Μάιερ, Σμιτ. Άλλος κανείς. Και φαινόμενος, λοιπόν, Βάιλερ, Σμιτ, Ρούλε, Μάιερ. Ποιος άλλος είπαμε. Αυτή. Σβάπ. Μάλιστα. Ωραία. Κυρία Βάιλερ, οι σκιώδεις εισηγητές είστε για σήμερα. Σας ορίζω σκιώδεις εισηγητές για σήμερα. Beide auch gleich weg, aber äh, es ist mir doch ein ναι. Θα πρέπει να τοποθετηθώ στο θέμα αυτό και θέλω να το πράξω, διότι θυμάμαι πολύ καλά ότι είχαμε στην προηγούμενη θητεία ένα πακέτο, μία δέσμη μέτρων που εγκρίναμε ομόφωνο μάλιστα σχεδόν εδώ στο Κοινοβούλιο, όπου καλούσαμε τα κράτη-μέλη επιτέλους και επιτέλους, ύστερα από 10 χρόνια τουλάχιστον παραγνώρισης των ευρωπαϊκών συνθήκων, να τηρήσουν το ευρωπαϊκό δίκαιο των συμβάσεων. Για τα θέματα των εξοπλισμών ξέρουμε ότι δεν είναι δημόσιες ε, οι συμβάσεις των προμηθειών, έστω το γνωρίζουμε, αλλά στην πράξη το 95% των συμβάσεων χαρακτηρίζονταν ως απόρριτες και μόνο το 5% μπορούσε να καταστεί δημόσια γνωστό. Εδώ πλέον αλλάζει η κατάσταση και γι' αυτό προτείνω και η και εσείς κύριε Πρόεδρε να ζητήσετε εξάπαντος από την Επιτροπή αλλά και από την Υπηρεσία Ευρωπαϊκή, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνα να σα κάνουν μια αναλυτική κατάσταση των σχετικών προμηθειών. Πριν από τι διακοπέ είχα ξεκινήσει αυτή την προσπάθεια επαφών και από ό,τι κατάλαβα το 1 τρίτο των κρατών μελών τουλάχιστον δεν έχει καν περάσει σε εφαρμογή το νομοθέτημα αυτό. Φαίνεται ότι δεν έχουν καν αντιληφθεί ότι υπάρχει αυτή η οδηγία και απλώ περιμένουν να δουν πού θα βγει η κατάσταση. Αυτά λοιπόν. Καταρχά μια μεγάλη κριτική για τον τρόπο τη συμπεριφορά απέναντι στο Κοινοβούλιο. Ε, τα άλλα δύο θεσμικά όργανα δεν έχουν τηρήσει τα όσα έχουν αποφασιστεί και βέβαια δεν τηρείται η προθεσμία για την μεταφορά σε εθνικό δίκαιο από ό,τι φαίνεται. Και δεύτερον, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να πω ότι δεν είναι τραγικό για μένα το να μην ενισχυθούν οι προπολογισμοί για την αμυντική αμυντικοί γιατί βλέπουμε ότι τουλάχιστον στη Γερμανία μια σειρά από ε, εικονικές αγορές, από καταχρήσεις, ανεξάρτητος του ποιος προκαλεί τι, ποιος κάνει ποια σύμβαση, που εν πάση περιπτώσει για 10 χρόνια τουλάχιστον πρέπει να περιμένουμε συχνά για να αποκαλυφθούν αυτές οι καταχρήσεις και ως ε, νεαρή Ω νεαρή πολιτικό θυμάμαι να έχουμε ξεκινήσει να, να εξετάζουμε ένα σκάνδαλο εξοπλισμών, το οποίο ακόμα τώρα αποκαλύπτεται σιγά σιγά. Ε, γι' αυτό λοιπόν νομίζω ότι θα ήταν καλό να διεκδικήσουμε μια σαφή και διαφανή διαδικασία και βέβαια πάντοτε έχοντας γνώμονα την ασφάλεια των στρατιωτών μας γιατί δεν συμβαίνει πάντα αυτό πρέπει να πω. Γίνονται αγορέ εξοπλισμών, ακριβών ή φθηνών δεν έχει σημασία, Χωρί όμως να λαμβάνεται μέρημνα για την ασφάλεια του στρατιωτικού προσωπικού που δραστηριοποιείται. Ε, αυτό πρέπει λοιπόν να αποτελέσει πρώτο και κύριο κριτήριο. Για τις ικανότητες, για τις επικρίσεις, τα ε, συμμερίζομαι τις ε, προτάσεις σας. Ε, χρόνια τώρα επισημαίνουμε τα ίδιες επικρίσεις και δεν βλέπουμε να έχει προχωρήσει η υπόθεση αυτή. Ήμουν, μάλιστα σκιώδη συγγήτρια στη μεγάλη συζήτηση που είχε γίνει στο παρελθόν. Δεν αρκεί να περιοριστούμε σε ένα ψήφισμα. Πρέπει να προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο γιατί όταν έχουμε αποφασίσει κάτι, όταν έχει κάτι εγγραφεί σε νομοθέτημα, το να μην εφαρμόζεται από το Συμβούλιο είναι παράδεκτο. Ευχαριστώ, έχετε δίκιο. Και εσείς νομίζω, κυρία Ρούλη, ήσασταν τότε εισηγείτε, έτσι δεν είναι, σας θυμάμαι. Ο κύριος Σμιτ, παρακαλώ. Μετά η κυρία Ρούλα. Ε. Um, Ευχαριστώ. Πολύ, καλή είναι, ε, πολύ καλό είναι το σχέδιο, δεν έχω πολλά να πω, όπως ε, ήταν και πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, αλλά είναι πολύ δέστος ο τομέας. Εγώ προέρχομαι από μικρή ουδέτερη χώρα, που εδώ και 200 χρόνια δεν έχει κάνει πόλεμο. Part of that, at least the... Αλλά τα τελευταία 15 χρόνια τουλάχιστον πιστεύαμε ότι αυτό οφείλεται στο ότι είναι ιδιαίτερα ε, κρατιά η βιομηχανία μας, η αμυντική μας βιομηχανία. Ε, και 80-90% ε, το εξάγουμε υποστηριζόμενοι από τους άλλους Αμερικανούς οποιονδήποτε. Και δεν μπορούμε να μην συζητήσουμε γενικότερα την αμυντική πολιτική και να συζητάμε ένα τέτοιο θέμα ε, για να είμαστε και ρεαλιστές. Είναι καλό να έχει η Ευρώπη αμυντική πολιτική. Κάποιοι αυτό πιστεύουν, εγώ πάλι όχι. Εγώ πιστεύω ότι είναι καλό να συμπαραταθούμε όλοι στο ΝΑΤΟ και να πείσουμε τον πρόεδρο Ομπάμα και τους Αμερικανούς να μην ε, ασχολούνται μόνο με τον ειρηνικό. Πρέπει να είναι γενικότερα ισχυρό το ΝΑΤΟ. Συμφωνώ με τους ε, γερουσιαστές. Ε, πήγα στο Κογκρέσο, συναντήθηκα με διάφορους και μου είπαν γιατί δεν πηγαίνετε εσείς. Ε, είδατε στη Λιβύη τι έγινε, ποια προβλήματα αντιμετωπίσαμε. έγιναν παραγγελίες για ελικόπτερα. Δεν έγινε τίποτα άλλο φοβερό. Δεν είμαι και ειδικό, αλλά πάντως για τη δική μας επιτροπή αυτό που πρέπει να μας απασχολεί είναι οι προμήθειες. Κρατικές προμήθειες. Δεν ξέρω αν υπάρχει ιδιαίτερο καταναλωτικό ενδιαφέρον για τα ελικόπτερα. Αλλά δεν μπορούμε να αποφύγουμε το βασικό ερώτημα τι είναι καλό για την Ευρώπη. Και ξαναλέω, εγώ δεν είμαι υπέρ της δημιουργίας Ευρωπαϊκού στρατού. Τέλο πάντων, είναι καλή αυτή η γνωμοδότηση, το ίδιο και η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Α μην είμαστε αφελείς, ε, ούτε φέτος θα το λύσουμε το πρόβλημα, πρόεδρο. το πλέον εύστοχο σχόλιο ήταν το τελευταίο που κάνατε, το πλέον εύστοχο δηλαδή της ε, χρονιάς. Κύριε ναι, συμφωνώ και εγώ. Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε πάντα με πολιτική αμυντική, αλλά με τις αρμοδιότητες. Και αυτό που δεν βλέπω μέσα στην έκθεση είναι η αναφορά σε υφιστάμενα νομοθετήματα στον τομέα αυτών που υφίστανται, που θα έπρεπε να εφαρμόζονται, γιατί εμεί έχουμε εγκρίνει νομοθέτημα στην Επιτροπή μα και θυμάμαι ότι ήταν αρκετά δύσκολα, γιατί ήμουν και εισηγήτρια ενό τμήματο σχετικού με τι μεταφορέ και, και θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό το ότι επιτύχαμε σύμβαση συμβαστική λύση και εγκρίναμε το σχετικό νομοθέτημα, το οποίο όμω τώρα δεν εφαρμόζεται. Είναι παράδεκτο αυτό και νομίζω ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε στην έκθεση αυτή, στην έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συμφωνώ με την κυρία Βάιλερ να ε, μεριμνήσει ώστε να τηρείται και να εφαρμόζεται σωστά η οδηγία αυτή στα κρατη Τίποτε παραπάνω. Όλα τα άλλα τα απορρίπτω είναι φιλοσοφικές τοποθετήσεις οι οποίες δεν προσφέρουν τίποτα σε εμάς εδώ στην Επιτροπή. Κύριε Σόμπερμαϊερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η έκθεση της Επιτροπής κινείται μεταξύ ε, καταγραφής της πραγματικότητας και έκφρασης ευσεβών πόθων, που δεν ξέρουμε και αν θα υλοποιηθούν. Πρέπει να δούμε βεβαίως τι αντιμετωπίζει η βιομηχανία, υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις σε συμβάσεις, δεν αναλαμβάνει νέα συμβόλαια ο κλάδος και γι' αυτό θα πρέπει να προσφέρουμε προτάσεις για μια ε, καλύτερη προστασία από την οικονομική κατάρρευση του κλάδου και όχι επιπλέον επιβάρυνση. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα πρόβλημα που αφορά τον κλάδο αλλά και την έλλειψη της οικονομικής υποστήριξης από τα κράτη-μέλη. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να δούμε σε ποιο βαθμό οι τεχνολογικές προδιαγραφές μπορούν να χαρακτηριστούν απόρριτες αλλά από την άλλη θα πρέπει να πω ότι όταν βλέπουμε στοχοθέτηση ε, Τη αξιοποίηση των χρονολογικών αυτών προδιαγραφών για λόγου παρακολούθησης. Δεν είμαι βέβαιος ότι καταλαβαίνω ακριβώς ποια είναι αυτή η στοχοθέτηση και τι επιδιώκεται. Οι δυνατότητες νομίζω θα πρέπει να εξεταστούν κατά τρόπο πρακτικό και πέραν τη νομολογίας βεβαίω. Η ανταγωνιστικότητα στον χώρο της άμυνας, της αμυντικής βιομηχανίας, ε, σημαίνει ποιότητα, σημαίνει προδιαγραφές, σημαίνει προϊόντα χρήσιμα, προϊόντα που μπορούν να πολιθούν σε πολλές ε, περιοχές του κόσμου, που μπορούν να προσφερθούν σε διαφορετικές αγορές και ως το δυνατόν μεγαλύτερα νούμερα με χαμηλότερο κόστος στην παραγωγή. Η ενίσχυση της διαφάνειας που βλέπω εδώ. Καλή μου ακούγεται, αλλά είναι δύσκολο ίσως να τηρηθεί, γιατί δεν έχουμε να κάνουμε θέματα απορρίτου. Η καινοτόμος ανάθεση συμβάσεων. Δεν μου φαίνεται ότι είναι πολύ καλός ο ορισμός, είναι λυπής, ασαφής, όσο καλή και αν είναι η ιδέα. Η αντιμετώπιση του υπερβολικής ικανότητας παραγωγής και των πλεονασμάτων ασφαλώς είναι μια λογική ε, απέτηση. Η υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η καλύτερη διασύνδεσή τους ασφαλώς είναι ενδιαφέρουσα πρόταση αλλά δεν είναι σαφώς διατυπωμένη. Ο χώρος πληροφορικής και των ηλεκτρονικών υπολογιστών ασφαλώς έχει πολύ μεγάλη σημασία και για το μέλλον. Καλή λοιπόν η προσέγγιση, καλές οι ιδέες. Ε, στις λεπτομέρειες όμως βλέπω ότι υπάρχουν σαφείς ελλείψεις. Είναι πολύ γενικόλογες δηλαδή οι περιγραφές. Μάλιστα. Κύριε Σπάπ, εσείς τώρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πολλά υπόθηκαν ήδη. Θα υπενθυμίσω πάντως ότι η Επιτροπή μας και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2008 με ε, εισηγητή τον κύριο Λάμπστορφ, τον συνάδελφο, είχαν στήσει τη συγκεκριμενοποίηση του άρθρου 296 της Συνθήκης για τη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με πολύ μεγάλη προσοχή υλοποίησαν, ε, ε, κατέγραψαν σε πρακτικούς όρους ε, το νόημα του άρθρου αυτού συμπεριλαμβάνοντας και προστατεύοντας και το εθνικό συμφέρον σε κάθε περίπτωση και δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην θεωρούνται σήμερα ακόμη επίκαιρες παρατηρήσεις ή ιδέες που είχαν διατυπωθεί τότε και να μην εφαρμόσετε το πλαίσιο αυτό της οδηγίας. Γι' αυτό λοιπόν η υλοποίηση του άρθρου 296 όπως είχε τότε σε συνδυασμό με την οδηγία του 2008 είναι ένα ζήτημα ακόμη επίκαιρο, ένα ζήτημα το οποίο έχει πολύ μεγάλη πολιτική σημασία όπως και παλιά. Θα υπενθυμίσω πάντως ότι το 2010, κύριε Πρόεδρε, αν έχετε την καλοσύνη, ίσως το μικρόφωνο σας θα ήταν καλό να το κλείσετε, τουλάχιστον, αν έχετε την καλοσύνη. Και θα ήθελα να πω λοιπόν ότι η Επιτροπή Άμυνας και Ασφάλειας είχε μιλήσει σε μια, έκθεση, σε μια μη νομοθετική έκθεση πρωτοβουλίας για τον περιορισμό της ικανότητας παραχωχής, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι επειδή έχουν περάσει τόσα χρόνια δεν είναι ακόμη επίκαιρο το αίτημα αυτό του νομοθέτη. Και όπως είπε η κυρία Ρούλα, πρέπει ακόμα τα κρατη να κληθούν να εφαρμόσουν την οδηγία που έχει εγκριθεί από το 2008. Εγώ είμαι διατεθειμένος να συζητήσω προσαρμογές και προποθέσει, αλλά επαναλαμβάνω ότι δεν έχουμε να κάνουμε δημόσιε προμήθειε, έχουμε να κάνουμε μια ευρωπαϊκή αγορά που αφορά ναι τα αμυντικά προϊόντα, τα προϊόντα τη αμυντική βιομηχανία, αλλά και η επαλήθευση τη οδηγία είναι αντικείμενο τη έκθεσή μα, και πρέπει να επενθυμίσουμε ότι και η έκθεση τη κυρία Ντίκο Καλπέ είχε πολύ σημαντικό έργο προσφέρει και θα πρέπει και αυτή να την αναφέρουμε. Ευχαριστώ. Ωραία, να πω και εγώ δύο πράγματα. Η κυρία Ρούλε πολύ σωστά ομίλησε όταν είπε ότι πρέπει να υλοποιηθούν οι ισχύουσε διατάξει βέβαια η όλη εξέλιξη στον τομέα των αμυντικών από τότε που ξαναργαζόμαστε πάνω σε αυτόν ε, χαρακτηρίστηκε από την ενοποίηση και τη συρρήκνωση όμως των αμυντικών προϋπολογισμών. Εξού και η αποτελεσματικότητα ε, των αγορών ε, εξοπλισμών ε, προσλαμβάνει μεγαλύτερη σημασία. Η Κομισιόν έχει εκπονήσει ένα πολύ καλό έγγραφο και σε ό,τι αφορά τη το, το, το αμυντικό τομέα είναι πάρα πολύ σημαντικό να επεξεργαστούμε καινοτόμε λύσει ε, σε ό,τι αφορά την ε, καινοτομία ε, για να διαφοροποιηθούμε και από το... μάλλον όπως έκαναν το 50 στην Αμερική. Το pre-commercial procurement είναι κάτι που φαίνεται ότι θα θελήσει να το υποστηρίξουν προγραμμάτες η Κομισιόν θα υποβάλω λοιπόν τροπολογίε ε, γιατί δεν πρέπει να αφήσουμε να χαθεί αυτή η ευκαιρία. Επίση, θα ήθελα να πω ότι οι βασικέ ε, μεταρρυθμίσει ε, του τομέα των δημοσίων συμβάσεων που μόλι εγκρίναμε πρέπει να εφαρμοστούν και στον αμυντικό τομέα το συντομότερο δυνατό, διότι ορισμένα από τα ζητήματα είναι να ενθαρρυντούμε τις ΜΜΕ και να υπάρχει μια προσέγγιση σε αμυντικές λύσεις όπου η ποιότητα της λύσης σε σχέση με, ε, την τιμή της ε, θα μπορούσε να αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό παράγοντα. επίση απλούστευση των διαδικασιών και διαθεσιμότητα ενός ε, καινοτόμου σχεδίου συνεργασίας στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων. Η άμυνα είναι άκρος ε, εξειδικευμένος τομέας. Θα μπορούσαμε λοιπόν ε, να ζητήσουμε την Κομισιόν ε, να εξετάσει συγκεκριμένα αυτό το θέμα της καινοτόμου, των καινοτόμων δημόσιων συμβάσεων. Θα μπορούσε να γίνει στον αμυντικό τομέα ένα πιλωτικό πρόγραμμα πάνω σε, αυτή, σε, αυτό, σε ένα καινοτόμο τέτοιο πρόγραμμα για τις δημοκρατίες στον τομέα των ε, δημοσίων συμβάσεων για την αμυντική βιομηχανία. Θα κάνω λοιπόν τροπολογίες και πιστεύω να συνεισφέρω στη σημαντική αυτή πρόταση. Τα πρότυπα ε, που είναι δική μας αρμοδιότητα αναφέρονται. Εμείς ε, θα ολοκληρώσουμε σύντομα την μεταρρύθμιση της όλης διαδικασίας για την κατάρτιση των προτύπων. Μιλάμε για κάποια υβριδικά πρότυπα ε, που θα μπορούσαν να έχουν ενδεχομένω και στρατιωτικέ εφαρμογέ. Είναι κάτι που δεν το είχα ξανά Αυτά τα υβριδικά πρότυπα, τέλο πάντων θα πρέπει να το εξετάσουμε. Και υπάρχουν και διάφορα άλλα αναλυτικά σημεία πάνω στα οποία θα πρέπει να ε, αναλύσουμε περισσότερο τα πράγματα. Θα ήθελα να πω ότι δεν υπάρχει ένα αντίγραφο ε, της Επιτροπής θέλουν βέβαια να εγκριθεί πριν από την άτυπη μάλλον όχι καθίστε να τα πω ανάποδα. Υπάρχει άτυπη επισκεψη, ε, μάλλον συνάντηση Υπουργών Άμυνα. Αυτή την ώρα μάλιστα στο Βίλνιους συνεδριάζουν και μετά θα έχουμε συζήτηση στο ευρωπαϊκό, στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφή το Δεκέμβριο. Το Κοινοβούλιο ε, έχει ένα στενό χρονοδιάγραμμα ακριβώ για να προλάβει αυτέ τι προθεσμίε. Θα δώσω το λόγο στην Κομισιόν. Αυτό που έχω να πω όμως είναι ότι είναι πολύ στενή η προθεσμία 12 Σεπτέμβρη λίγη για την κατάσταση τροπολογιών και θα ήθελα να σας παρακαλέσω ή δυνατόν να υποβάλλετε στα αγγλικά της τροπολογίας σας λόγω ακριβώς του λιγού διαθέσιμου χρόνου. Πραγματικά πρέπει να ψηφίσουμε στην ΜΜΚΟ στις 30 Σεπτεμβρίου για να μπορέσει η Επιτροπή ε, η αρμόδια να ολοκληρώσει την έκθεσή της πριν από τις 26 Οκτωβρίου που θα τεθεί το θέμα στη διάσκεψη κορυφής. Αυτά είχα να πω εγώ. Υπάρχει κάποιος άλλος που θα ήθελε το λόγο. Αν όχι, να δώσω το λόγο στην κυρία Κατσιούμπερς. Λίγα λεπτά μόνο έχετε στη δεσία γιατί μας τελειώνει ο χρόνος. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι πάρα πάρα πάρα πολύ σύντομη. Συνολικά Μα ικανοποιεί πολύ το σχέδιο γνωμοδότησης με την παρούσα του μορφή. Δεν έχουμε λοιπόν κάποιο σημαντικό σχόλιο πάνω στο περιεχόμενο της γνωμοδότησης, αλλά θα ήθελα να σχολιάσω ορισμένε από τις παρεμβάσεις. Πρώτα απ' όλα, σημειώνω ότι η ενίσχυση της ενιαία αγορά στον τομέα της άμυνας και αμυντικέ αγορέ ήταν, η αμυντική αγορά μάλλον ήταν και μια από στην ανακοίνωσή μα. Γι' αυτό και χαιρόμαστε που βλέπουμε την ισχυρή υποστήριξή σα και στην ανακοίνωση. επίση λέγαμε ότι πρωταρχικό στόχο εδώ είναι η υλοποίηση τη νομοθεσία που έχει εγκριθεί μέχρι τώρα. Και συγκεκριμένα εγκρίθηκε πριν από λίγα χρόνια. Εξ όσων γνωρίζω, για να προσθέσω κάτι, δεν τα πάμε και τόσο κακά με την ε, με, μεταφορά της ε, δημοθέσης αυτής του εθνικό δίκαιο σε ό,τι αφορά την οδηγία για τις δημόσιες προμήθειες τουλάχιστον μέχρι τώρα όλα τα κρατημέλη, εξ όσων γνωρίζω παλαιβάνω, την έχουν ε, μεταφέρει στο εθνικό δίκαιο. Αυτό το οποίο προτείνουμε όμως είναι ανακοίνωση, είναι και στο πλαίσιο της δράσης που λέγεται να παρακολουθήσουμε το άνοιγμα των αμυντικών αγορών των κρατών μελών, τι σημαίνει αυτό, σημαίνει ότι θα παρακολουθούμε ε, σε τακτά διαστήματα τις χρηστές νομοθετικές πρακτικές, ε, την ε, υλοποίηση της νομοθεσίας που έχει προταθεί και έχει εγκριθεί και από το Κοινοβούλιο. Αυτό θα γίνει ως προς αυτό το κομμάτι. Επίσης, σε ό,τι αφορά το pre-commercial procurement, είναι ένα ενδιαφέρον εργαλείο, σας ευχαριστώ που το αναφέρατε και χαιρόμαστε που υπάρχει υποστήριξη ε, να γίνει μνήα ε, του στην γνωμοδότηση. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρος, δεν απαντήσατε όμως αν αυτό το καινοτόμο, το, το, εργαλείο της καινοτόμου, καινοτόμων διαγωνισμού, θα μπορούσατε να το χρησιμοποιήσετε και να φτιάξετε ένα πιλωτικό πρόγραμμα σχετικά Τέλο πάντων, α συμφωνήσουμε πρώτα σε επιτροπή να του περιλάβουμε και μετά μπορείτε να μα πείτε την άποψή σα. Να δώσω το λόγο στην συγκεκριτή για να ολοκληρώσει. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλου του συναντέλου για τι παρατηρήσει, τι υποδείξει. Ήταν άκρως ενδιαφέροντα όλα τα σχόλια, Όπω ανέφερε και ο πρόεδρο. Είναι πάρα πολύ στενό το χρονοδιάγραμμα, πάρα πολύ μικρές προθεσμίες. Γι' αυτό Έπρεπε να ξεκαθαρίσουμε τι είναι αρμοδιότητα της ΙΤΡΕ, τι είναι αρμοδιότητα της ΙΜΚΟ. Έπρεπε να χαράξουμε αυτή τη διαχωριστική γραμμή τώρα. Αυτό έχει γίνει, γνωρίζουμε ποιο είναι το δικό μας πεδίο αρμοδιότητας και έτσι μπορούμε να καταλήξουμε στη δική μας γνωμοδότηση. Για παράδειγμα, η οδηγία για την μεταφορά μυντικών προϊόντων εντάσσεται στο πεδίο αρμοδιότητας της ΙΤΡΕ, εξού και δεν έκανα λόγο για το συγκεκριμένο θέμα. Άκουσα με προσοχή όλες σας τις υποδείξεις και συστάσεις ε, και συμφωνώ με το μεγαλύτερο μέρος των παρατηρήσεων των συναδέλφων, οι περισσότεροι από τους οποίους μίλησαν για το πόσο σημαντικό ήταν το γεγονός ότι ακούστηκε η φωνή του Κοινοβουλίου, το οποίο κατέληξε σε μια ξεκάθαρη θέση. Εξέφρασε δηλαδή την προτίμησή του σε, στις καινοτόμες πρακτικές στις δημόσιες συμβάσεις. Οι δημόσιες συμβάσεις σίγουρα είναι ένας τομέας που χρειάζεται μια αναβάθμιση, μια βελτίωση. Η κανόνα εμπιστευτικότητα σε απορρίτω χημίκες πρέπει να αναθεωρηθούν. Έρχομαι τώρα στις ΜΜΕ, όχι μόνο γιατί τις αγαπώ πάρα πολύ, αλλά και γιατί η επίθεση μου αποτελεί ότι με το ευρωπαϊκό κλάστερ της στάδες επιχειρήσεων και τις καινοτόμες αυτές στάδες επιχειρήσεων θα μπορούσε ε, να γίνει μεγαλύτερη συμβολή των ΜΜΕ στον τομέα αυτό, που δεν είναι μόνο πρώτος κρίκος ε, στην αλυσίδα εφοδιασμού. Μάλλον να μην γίνουν ο πρώτος κρίκος, αλλά τέλος πάντων να μπουν σε αυτή τη διαδικασία η αμυντική βιομηχανία δεν είναι πλέον, δεν έχει να κάνει με εξοπλισμούς παλιά σχολής. Πάει αυτό. Μιλάμε τώρα για καινοτόμες λύσεις, για απάντηση σε περιφερειακές διανέξεις, σε καινοτομίες καινούργιες, νεωτερικές. Ορισμένα κράτη-μέλη μπορεί να μην είναι έτοιμα για κάτι τέτοιο ή υπάρχει και σπάνιση πόρων, ένα άλλο παράδειγμα. Λοιπόν, δεν έχουμε πολύ χρόνο, όπως είπα, ε, είναι πολύ σαν το χρονοδιάγραμμα. 12 Σεπτεμβρίου, παρακαλώ, το αργότερο να έχω λάβει τις τροπολογίες σας. Ε, πρόεδρος, ευχαριστώ και επαναλαμβάνω στα αγγλικά ή δυνατόν τροπολογίες. Ευχαριστώ και την εκπρόσωπο της Κομισιόν. Θα περάσω τώρα στην έκθεση του κυρίου De Jongs, δεύτερη έκθεση De Jong για σήμερα για τις πρακτικές παραπλανητικής διαφήμισης. εξέτας τροπολογιών. Ξέρω ότι έχετε κάνει μεγάλη περίοδο, 54 συντροπολογίες, αλλά έχουμε και 6 συμβαστικές τροπολογίες που θα συζητήσουμε. Όλοι οι σκιώδεις νομίζω είναι παρόντες, ΦΑΠ, Πρέντεργκάστ, Ροσφόρ, Ρούλε, Μπίλαν. Όλοι είναι εδώ. Λοιπόν, θα σας παρα καλέσω να παρουσιάσετε εσείς τις τροπολογίες. Και ο κύριος Πέτρη είναι εδώ. Πολύ τακτικός επισκέπτης και παλιός φίλος, θα έλεγα, της Επιτροπής μας. Και έχουμε και το τελευταίο θέμα ε, το... του κύριου Σφάπ. Λοιπόν, ο Ντένις έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ. Έχετε και τις συμβαστικές τροπολογίες. Μπορώ να σας πω ότι με μεγάλη χαρά ασχολήθηκα με αυτό, διότι ήταν όλες οι τροπολογίες επικοδομητικές και έτσι ε, ενισχύεται και το περιεχόμενο της έκθεσης. Πέρα από αυτά τα έγγραφα που έχετε, όλοι οι σκιώδεις, όπως και εγώ, λάβαμε ένα mail από τον Ανδρέα Σουάμπ, που πέρα από αυτά που λέει για τις συμβαστικές και κάνει και προτάσεις που, με τις οποίες δεν έχω κανένα πρόβλημα, κάνει και μια πρόταση για μια συμβαστική τροπολογία για το εκτιμώντας α και Πιστεύω ότι είναι καλή ιδέα. Βλέπω τις λεπτομέρειες, συγκρίνω τι τροπολογίε και τέλο πάντων δεν είδα και πολύ χρόνο στη διάθεσή μου. Πριν από τη συνεδρίαση το πήρα το mail, αλλά εκ πρώτης όψεως μου φαίνεται ότι θα τα καταφέρουμε, θα συμβαστούμε. Κύριο Σφαντ. Πρόεδρε, έχω καταθέσει γραπτός τις προτάσεις. Έχω λάβει μάλλον γραπτός Έχω αποστείλει γραπτό στις προτάσεις στους συναδέλφους. Νομίζω ότι αρκεί, δεν χρειάζεται να συζητήσουμε. Χαίρομαι που ο κύριος Διόγκ ενδιαφέρεται και συμβάλλει. Πολύ ευχαριστώ στο λάβω υπόψη τις προτάσεις που θα κατευθούν. Ευχαριστώ. Thank you very much, Mrs. Prendergast. Ευχαριστούμε κύριε Prendergast. Ε, ευχαριστώ. Ε, θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Ντεγιόν καθώς και τους υπόλοιπους συναδέλφους που ασχολήθηκαν με το φάκελο, κυρίως για το επαναλαμβανόμενο πρόβλημα που έχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έχουν ένα σημασιολογικό ζήτημα με τη συμβαστική 2. Μου φαίνεται ότι είναι δυσανάλογο να αναφερόμαστε σε προμήθευτες υπηρεσιών και να τους χαρακτηρίζουμε enablers, ε, δηλαδή ε, ε, τους αποδίδονται δραστηριότητες που δεν αναλαμβάνουν. Πιστεύω λοιπόν, ελπίζω ότι ο κύριος Ντε και οι συνάδελφοι θα επανεξετάσουν ε, την ε, διατύπωση που προτείνω για την 29 και καλό θα ήταν να εξετάσουμε και το ενδεχόμενο να εισαγάγουμε ε, υποχρεώσεις για τους οργανισμούς σχετικά με τις παραπλανητικές πρακτικές, οπότε η συμβαστική 5 είναι μία που μπορούμε να υποστηρίξουμε αν ψηφίσουμε την 46 ξεχωριστά. Συμβαστικές 1, 2, 3 και 4 επίσης μας βρίσκουν σύμφωνος. Είχα εκφράσει ενδιασμούς για τη συμβαστική 3, αλλά πιστεύω ότι η τροπολογία 1 τώρα τις ανησυχίες μας για τη συμβαστική 6. Δεν είμαι πεπισμένη ότι η τροπολογία 52, το πνεύμα της τροπολογίας 52 που είχα καταθέσει έχει ενσωματωθεί. Ε, μιλάμε για ε, ιδιωτικές λύσεις ε, εφαρμογής ε, σε επίπεδο κρατών μελών όπως στη Γερμανία που κάποιες ενώσεις αναλαμβάνουν δραστηριότητες που υπερβαίνουν το πεδίο της συλλογική αποζημίωσης. Δηλαδή θέλω να διευρύνουμε το πεδίο εφαρμογής. Σας ευχαριστώ και πάλι. Ευχαριστώ τον κύριο Ντεγιάν και τους συναδέλφου. Σας ευχαριστούμε εμείς, κύριος Γοσφό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ντεγιόγκ Όπω και οι συνάδελφοι, είναι πολύ επικοδομητικό ο τρόπο που δουλεύει γιατί λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσει μα. Στην ε, συμβαστική τροπολογία 1 είχα κάνει παρατηρήσεις διότι φοβόμουν ότι στιγματίζεται τις επιχειρήσεις ο μαύρος κατάλογος. Όμως ο μαύρος κατάλογος των ε, αθέμητων εμπορικών πρακτικών είναι μια πολύ καλύτερη λύση διότι όταν υπάρχουν κατά να πάτε για τις εταιρείες μπορούν να καταχωρηθούν σε αυτό τον κατάλογο και μπορούμε να συμφωνήσουμε πλέον με αυτό το μαύρο κατάλογο. Τώρα για τη συμβαστική, για την παράγραφο 11 έχω ένα ερώτημα. Θυμάστε ότι αναφερόμαστε εδώ ε, στην αλλαγή του πεδίου εφαρμογή για να καλύπτει και το B2B, γιατί προ το παρόν ε, περιορίζεται στι σχέσει τη επιχειρήσεων με του καταναλωτέ. B2C. Το Κοινοβούλιο είχε ζητήσει την Επιτροπή να κάνει μια σχετική πρόταση. Δεν νομίζω να συμβεί αυτό, γιατί όπω ξέρετε ε, τώρα επεξεργάζονται μια διαφορετική οδηγία για αυτό το ζήτημα, άρα οι σκιώδεις πρέπει να επανεξετάσουν αυτό το θέμα της συμβαστικής ε, τρία που αναφέρεται στην παράγραφο 11, διότι δεν είμαι πλήρως ικανοποιημένος. Για την συμβαστική 2 Εκεί λέμε ότι οι τράπεζες, οι τηλεφωνικές εταιρείες πρέπει να υπομισθούν με διαφορετικό τρόπο τις ευθύνες τους. Συμφωνώ να είναι λίγο πιο ήπια η διατύπωση. και για τις ε, συλλογικές προσφυγές και για την εκπροσώπηση των θυμάτων, θέμα κέρια σημασίας για την ομάδα μου, ε, θα θυμάστε ότι υπήρχαν κάποια ερωτηματικά και τώρα θυμίζω ότι στα κράτη-μέλη στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται η δυνατότητα ε, κίνησης συλλογικών αγωγών ε, αυτό καλύπτεται πλέον στην τροπολογία και πάλι εδώ ακολουθούμε τη σωστή κατεύθυνση. Δεν θέλω να δεσμευτώ ήδη σήμερα, αλλά κατά πάσα πιθανότητα θα μπορέσουμε να την υποστηρίξουμε. Ε, είναι αγαστή συνεργασία ε, εν γέννη και πολύ γρήγορα περάσαμε από το στάδιο της κατάστασης των τροπολογιών στην εκπόνηση των συμβαστικών τροπολογιών, οπότε εργαστήκαμε με άριστο τρόπο και μας συγχαίρω. Σας ευχαριστούμε κύριε Γοσφόγ, κυρία Ρούλε. Ναι, συμφωνώ. Και θα συζητήσουμε τις συμβαστικές τροπολογίες. Απλώς μια παρατήρηση για τον κύριο Ροσφόρ. Το B2B είναι μια πρόταση από την κυρία Wallace, δική σας συνάδελφο, από την δική σας ομάδα που έχει στήσει την επέκταση. Αυτό ήθελα να επισημάνω ότι προέρχεται από τους φιλελευθέρους. Μα αυτό είναι το, το πρόβλημα, ότι έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους με εμπειρία, αλλά η μνήμη μας είναι επιλεκτική. Κύριε Βίλα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω καταθέσει προς ε, προτάσεις μου Ορίστομαι λοιπόν στα πιο σημαντικά θέματα και θα ήθελα να επισημάνω στον Πρόεδρο ότι κάποιες εκ των τροπολογιών δεν ήταν αρκετά ακριβείς. Χρειάστηκε δηλαδή να αγνοήσω την πολιτική μετάφραση και να κοιτάξω το αρχικό κείμενο για να καταλάβω. Για τις ε, τροπολογίες υπάρχουν πιστεύω κάποιες που μπορούν να διατυπωθούν συμβαστικά γιατί υπάρχουν συναφείς με τις δικές μου 26, 25 βλέπω ότι βαίνουν προς την ίδια κατεύθυνση και μπορούμε να βρούμε ε, μία λύση με μία συμπίληση πρακτικών αθέμητων. Ξέρουμε ότι μπορεί να δημοσιοποιηθεί το όνομα κάποιου επιχειρηματία, κάποιου καταστηματάρχη, ο οποίος ε, ε, ακολουθεί αθέμητες πρακτικές, μόνο εφόσον ε, προηγηθεί απόφαση δικαστηρίου. Ε, αυτό θα πρέπει ίσως να το δούμε. Εγώ είμαι κατά της ε, κατάρτισης καταλόγου, μα, μαύρο πίνακα όπως τα λέγαμε, επιχειρηματιών για δε τις παραπλανητικές ε, πρακτικές. Θα προτιμούσα να μην επεκταθεί η οδηγία στο B2B, business to business. Για το 2015 θα πρέπει να γίνει λόγος και για το ρόλο των επιχειρήσεων που προσφέρουν συλλογικές υπηρεσίες. Οι επιχειρήσεις αυτά, οι συμφωνίες μπορεί μερικές φορές να οδηγούν σε παραπλάνηση. Δεν ξέρω όμως εάν μπορούν να θεωρηθούν παράνομες. Το παράνομο λοιπόν, τη λέξη παράνομες, ίσως θα πρέπει να τη διαγράψουμε και να ζητήσουμε περισσότερο έλεγχο στις δραστηριότητες των επιχειρήσεων. Για το άρθρο 46 δεν ξέρω χρειάζεται περισσότερο κανονισμή. Για το 16 θα προτιμούσαμε την θελοντική συμμετοχή, opt-in και την εξέταση των εγχώρων συστημάτων. Τροπολογία 51 που έχω καταθέσει εδώ, μου αρέσει καλύτερα. Στο 27 δεν έχω καταθέσει τροπολογία, αλλά η λέξη επιτρέπει, enables, νομίζω θα πρέπει να αντικατασταθεί από τη φράση υπάρχει των οποίων χρησιμοποιούνται οι υπηρεσίες». Είναι πολύ πιο ακριβής η διατύπωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους κοιόδης συγκητές. Σημειώνει ασφαλώς ο εισηγητής ε, της ε, παρεμβάσης σας. Κύριος Πέτρη, αν δεν θέλουν άλλοι συνάδελφοι, ας κάνει ένα σχόλιο. Και ιδιαίτερα για τα ένδικα μέσα που προβλέπονται να μας πείτε ποια είναι η γνώμη σας και μετά θα ακούσουμε τον εισηγητή. Κύριε Πέτρη. Ευχαριστώ. Όντως. Μπορούμε σε γενικές γραμμές να υποστηρίξουμε το σχέδιο του εισηγητή. Πιστεύουμε δε πως πολλές τροπολογίες ακολουθούν τη σωστή κατεύθυνση. Κυρίως δε οι συμβαστικές τροπολογίες που μπορούμε να υποστηρίξουμε εκτός από την υπαριθμόν 5 σε σχέση με τους οργανισμούς ίσπραξης οφειλών. Διότι αυτοί οι οργανισμοί δεν είναι σε θέση να εκτιμήσουν αν είναι παραπλανητικές οι πρακτικές πρωτού γίνει η πώληση. Οπότε προτιμούμε να παραμείνει ως έχει παράγραφος για την συμβαστική 3 για την πιθανή ε, διεύρυνση του πεδίου εφαρμογή οδηγία περί αθέμητων εμπορικών πρακτικών. Δεν συμφωνούμε με τη σχετική παράγραφο της έκθεσής σας και άρα καλωσορίζουμε την αλλαγή που προτείνεται συμβαστική τροπολογία ή ε, την τροπολογία 37 ως εναλλακτική λύση. Είναι ξεκάθαρο για την Επιτροπή ότι η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογή οδηγίε για τι αθέμητε πρακτικέ δεν είναι κάτι που μπορούμε να εξετάσουμε αυτή τη στιγμή, διότι υπάρχει ε, και σχετική έκθεση για την οδηγία B2C, οπότε... Όντως, μπορούμε να ασχοληθούμε ε, με ενδεχόμενη αναθεώρηση της σχετικής οδηγίας, αλλά τα προσεχή έτη, όχι αυτή τη στιγμή. Ε, συμβαστική έξι. τώρα μπορούμε να την υποστηρίξουμε πλήρως διότι ακολουθεί την πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις συλλογικέ αποζημιώσεις ε, ακολουθώντας και τις πρόσφατες για αυτό το ζήτημα συστάσεις. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ο Ντένις Γιόγκ για να συνοψίσει ίσως ε, και να κάνει κάποια σχόλια προετοιμάζοντας έτσι και την ψηφοφορία. Ευχαριστώ Μάλκομ. Ε, δεν θα ήθελα τώρα να σχολιάσω ξεχωριστά κάθε παρατήρηση που ακούσαμε. Νομίζω ότι γενικά ακολουθούμε όλη την ίδια ρότα. Ω προ αυτά που μα είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη σύσταση του Κοινοβουλίου για πιθανή διεύρυνση του πεδίου εφαρμογή οδηγία για τι αθέμητε εμπορικέ πρακτικέ, ε, είναι δύσκολο το Κοινοβούλιο να αποστασιοποιηθεί από αυτά που έχει ήδη αποφασίσει στο παρελθόν. Αυτή η συμβαστική τροπολογία είναι όντως συμβαστική και άρα ζητά μόνο αναθεώρηση. Και μας λέει η Επιτροπή ότι ούτως ή άλλως σκοπεύει να το κάνει. Αυτό ακριβώς ζητάμε μέσα στη συμβαστική τροπολογία. Εν ευθέτω χρόνο να γίνει αναθεώρηση. Ε, Μπορείτε νομίζω να κάνετε μια υποχώρηση σε αυτό. Τώρα για τις υπόλοιπες θα ήθελα να προτείνω το εξής. Ο κύριος Φάμ ε, μας βοήθησε πάρα πολύ γιατί έστειλε αυτά τα λεπτομερή σχόλια με email και είναι πολύ εύκολο για μένα έτσι να ε, προσαρμόσω τις συμβαστικές τροπολογίες ε, και θα ήθελα απευθυνόμενο στην κυρία Πέντελγκας και στον κύριο Χοσφόχ να ζητήσω να κάνω ακριβώς το ίδιο ένα email με συγκεκριμένες προτάσεις ε, για τις συμβαστικές τροπολογίες και ο κύριος Μπίλαν φυσικά. Αν και σε αυτή την περίπτωση νομίζω ότι η διάσταση απόψεων θα είναι μεγαλύτερη ε, σε σχέση με τους δύο υπόλοιπους, ε, τους δύο άλλους σκιώδους εισηγητές. Ας μου στείλετε ένα email και μετά το Στρασβούργο μπορούμε να κάνουμε μία σύντομη συσκέψη και να καταλήξουμε στο τελικό σετ συμβαστικών τροπολογιών. Πάντως είμαι αισιόδοξο. Νομίζω θα τα ρυθμίσουμε τα εκκρεμή ζητήματα. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και τους σκιώδες εισηγητές και όλους όσους ε, ήρθαν. Είχαμε πληρότητα απαρτίας και οδών για πέμπτη απόγευμα δεν είναι σύνηθες και δείχνει πόσο ενδιαφέρον είναι το θέμα. Περνάμε τώρα στο τελευταίο σημείο για σήμερα. Είναι μια πολύ σημαντική έκθεση του Ανδρέα Σφάπα για ένα πακέτο από την πλευρά Κομισιόν που έχει ως στόχο την εξασφάλιση κοινού υψηλού επίπεδου ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση. Ο Τζέπα Λαμόντι ανανεωμένος ε, ε βρίσκεται εδώ, εκπρόσωπος της Κομισιόν, αλλά από σκιώδης χωλένουμε. Έναν έχουμε μόνο. Δεν ξέρω, είναι εδώ κυρία Ρούλε, αλλά δεν είναι αυτή η σκιώδησε. Mm. Χαμόν Μέντες. So I think it may well be a between Mr. Schwab and myself. Άρα εγώ και ο κύριος Σβάμπ μόνο είμαστε ως ο Τέλος πάντων, έχω επίσης να κάνω ε, και κάποιες σοβαρές ανακοινώσεις για την ε, συμμετοχή άλλων επιτροπών. Ε, νέα είδηση έφτασε σήμερα, δεν ξέρω αν θέλει ο Αντρέας να πει κάτι. Λοιπόν, να σας επενθυμίσω καταρχάς εγώ που βρισκόμαστε, δεν ξέρω ούτε κι αν η Κομισιόν έχει ενημερωθεί σχετικά. Όπως γνωρίζετε, αυτό το πακέτο ε, μας ανατέθηκε από τη διάσκεψη των Προέδρων ώστε να είμαστε καθήλυνα αρμόδιοι. Όμως μια άλλη επιτροπή ε, αμφισβήτησε που δεν το δέχτηκε η διάσκεψη των Προέδρων. Εμείς είμαστε η, η καθήλυνα αρμόδια επιτροπή η Επιτροπή όμως, ε, η βιομηχανίας, ε, ήθελε να συμμετέχει δυνάμει του κανόνα 5, ε, να έχουμε δηλαδή διέρηση αρμοδιοτήτων. Αυτό συμφωνήθηκε τώρα. Η Επιτροπή τώρα πολιτικών ελευθεριών επίσης ήθελε να συνδεθεί, να συμμετάσχει. Με βάση τον κανόνα 49 συν. Δηλαδή να, καλεί, να καλείται ο εισηγητή του ε, και ε, να ενημερώνεται. Δεν συμφωνούσαν, θέλαν όμως μεγαλύτερη συμμετοχή. Ο κύριος Λένε, ο πρόεδρος Επιτροπής, ε, που έλεγε να μην το δεχτούν, η δέσκεψη των πρόεδρων δέχτηκε τη σύνδεση, αλλά με βάση τον κανόνα 50. Άρα θα έχουμε κάποια ζητήματα σε ό,τι αφορά τη διάκριση αρμοδιοτήτων. Τώρα δεν ξέρω με ποια βάση αυτή η απόφαση λήφθη από τη διάσκεψη των Προέδρων, δεν είμαι σίγουρος. Κάποιες φορές έτσι συμπεριφέρεται πάντως η διάσκεψη των Προέδρων. Είναι λίγο λοιπόν δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεται πλέον, ε, πλέον ο κύριος Φαπ. Επίσης, ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα, πρέπει να δούμε ακριβώς πώς θα μπορέσει να γίνει η πράξη αυτή η συνεργασία μεταξύ των επιτροπών θα μας τα πει ίσως καλύτερα ο κύριος Φαπ. Θα μας πει βέβαια και οτιδήποτε άλλο θέλει να πει, αλλά είναι η πρώτη εξέταση εκθεσή σας κύριε Φαμπ οπότε θέλουμε να δούμε και τι τροπολογίες προτείνετε για το σημαντικό αυτό θέμα. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob ich es ganz so σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δεν ξέρω βέβαια αν θα μπορέσω να είμαι τόσο απλός όσο ήταν ο κύριος Ντεγιόν. θα προσπαθήσω. Ε, ήθελα να του κάνω κοπλιμέντο. Τέλο πάντων, δεν τον βλέπω, έφυγε. Δεν μπορώ να μιλήσω ξανά με τον Σοσιοδόν εισηγητών. Με τον Ραμόν, ε, ε, τον σκιώδηση των σοσιαλιστών, έχω συνεργαστεί, μου ζήτησε να, γίνει, να αναβληθεί η υπόθεση με Δεν έχω πρόβλημα, μπορούμε να την αναβάλουμε για τις 24 Σεπτεμβρίου χωρίς πρόβλημα. Δεν μας δημιουργεί αυτό πρόβλημα για τη συνέχεια των συζητήσεων. Α, μέχρι και 1 Οκτωβρίου θα μπορούσαμε να πούμε. Λοιπόν, για μένα και για συναδέλφους από άλλες ε, επιτροπές συνταξή εκθέσεων, ξέρετε δεν είναι εύκολο να λειτουργήσουμε όταν δεν ξέρουμε πότε θα είναι έτοιμες οι εκθέσεις. Είμαστε στο τέλος της θητείας, 24 Σεπτεμβρίου. Δεν μου δημιουργεί πρόβλημα. Δεν νομίζω ότι θα κινδυνεύαμε να μην έχουμε ολοκληρώσει την έκθεση εντός των προθεσμιών. Είναι σαφές το χρονοδιάγραμμα λοιπόν. Θέλουμε να προσπαθήσουμε να ψηφίσουμε όσο ε, πριν λήξει η θητεία. Μέσα σε αυτό το έτος η Επιτροπή Ήτρε με την οποία είμαστε σε ενισχυμένη συνεργασία με, τον με την κυρία Ντελκαστήγιο. Εγώ έχω εξαιρετικέ επαφέ με την κυρία Ντελκαστήγιο. Προσπαθεί η ίδια να κάνει ό,τι μπορεί για να ψηφίσουν εκεί πριν από εμά. Ούτε η συμμετοχή της ΛΥΜΠΕ θα μας κάνει να χάσουμε χρόνο. Μιλάμε απλά για κοινέ αρμοδιότητες. Ουσιαστικά δεν θα είναι ε, σημαντική συμβουλή παρά μόνο σε, για ένα σκέλος της έκθεσης. Να έρθω τώρα στην ουσία κύριε Πρόεδρε. Ψηφιακό θεματολόγιο προβλέπεται το ενδεχόμενο διαταραχών λόγω, ε, μάλλον στο σύστημα μια χώρα θα μπορούσαν να επηρεάσουν ε, τι άλλε χώρε. Γι' αυτό είναι σημαντικό και δεν νομίζω ότι είναι αντίθετο κανεί προ αυτό. Είναι απαραίτητο να έχουμε σταθερές ε, διαδικασίες για να παράσχουμε εγγυημένες βασικές υπηρεσίες για την επέκταση της ψηφιακής αγοράς. Υπάρχουν διαφορετικοί κανόνες στην Ένωση. Προσπαθούμε να Έχουμε μια αναρμόνιση των προσεγγίσεων. Έχει κάνει μια εξαιρετική πρόταση κομισιών για τη δημιουργία συνθήκων που θα εγγυώνται μια σχετικά ομοιόμορφη ασφάλεια ε, δικτύων και πληροφοριών. Πρέπει να είναι ασφαλή τα δίκτυα για να μπορέσουμε να έχουμε μια καλή λειτουργία της κοινωνίας και της οικονομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά αυτό πρέπει να το διαχωρίσουμε από άλλους πολιτικούς ε, στόχους, προστασία δεδομένων, ε, τρομοκρατία, υπηρεσίες, ε, ποινικές διώξεις. Και έτσι μπορεί ε, να υπάρξει μια προσπάθεια για συγκάλυψη εγκληματικών δραστηριοτήτων και εμείς προσπαθούμε στο επίπεδο αυτό να μιλήσουμε για μια επίθεση για, ε, στην ε, ασφάλεια των δικτύων. Αυτό προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε, να αντιμετωπίσουμε καλύτερα. Εδώ λοιπόν δεν θέλουμε να το ανακατέψουμε το θέμα της προστασίας των δεδομένων. Δεν θέλουμε να αμφισβητήσουμε τίποτε σχετικό με τις αρμοδιότητες των διοκτικών αρχών, γιατί είναι θέματα των κρατών μελών. Απλώς ζητήματα που σχετίζονται άμεσα και δεσμευτικά με την εσωτερική αγορά και την ασφάλεια των δικτύων και των δομών, εκεί δηλαδή που μπορούν να υπάρχουν τέτοιου είδου κίνδυνοι, μόνο αυτά θέλουμε να συζητήσουμε. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ενισχύσουν το επίπεδο της άμυνας τους κατά τέτοιων επιθέσεων, λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και να προχωρήσουν σε συνεργασίες μεταξύ τους. Σε επίπεδο κρατών μελών, λοιπόν, σε επίπεδο Συμβουλίου, το συμπίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να ενταχθούν οι άμυνες αυτές, οι δυνατότητες άμυνες, άμυνας και αντιμετώπιση επιθέσεων στις ευρωπαϊκές δομές για να αντιμετωπιστούν και να επιληθούν και οι συγκρούσεις ε, και τα κενά. Η ε, κατανόηση των ε, κινδύνων για την ασφάλεια, τα ζητήματα της αντιμετώπισης, της αντοχής της απόκρουσης, επιθέσεων και ο αποκλεισμός βέβαια των μακροπόθεσμων βλαβών στις υποδομές. Και στόχος είναι η εξασφάλιση μιας ε, γενικότερης ασφάλειας των δικτύων με δεδομένη και την ανάγκη για ρύθμιση. Έχουμε θεσμικές δομές που μπορούν να ε, αξιοποιηθούν για την προστασία, την κυβερνοάμυνα όπως το λέγαμε και την ανάπτυξη μιας ανταλλαγής ε, γνώσεων, ε, πληροφοριών και το καθεξής μεταξύ θεσμικών και ιδιωτών, θεσμικών φορέων και ιδιωτών στα θέματα άμυνας και η διαχείριση κινδύνου βεβαίω από τους παρόχους θα πρέπει να ενισχυθεί. Και φτάνω στα τελευταία σημεία που θα ήθελα να θίξω κύριε Πρόεδρε, ότι η οδηγία στοχεύει στην εξασφάλιση για τις δημόσιες αρχές, βέβαια μέσα από ένα δίκτυο ε, επικοινωνίας της δυνατότητας για πλήρη ανταλλαγή πληροφοριών και ε, εμπειριών μεταξύ των κρατών μελών και την ε, απόκρουση κινδύνων για κρίσιμη σημασία υποδομών ώστε να υπάρχει και, και ταυτόχρονα να υπάρχει καλύτερη επισκόπηση την Ευρώπη για το ποιοι είναι οι κίνδυνοι και πώς μπορούν να προστατευτούν αυτές οι υποδομές. Η συζήτηση για την παρακολούθηση τη ε, παρακολουθήσεις, το NSA, το πρόγραμμα PRISM, έχει βέβαια σε ένα βαθμό το ρόλο του να παίξει. Στη Γερμανία αλλά και σε άλλα κράτη-μέλη οι συζητήσει δείχνουν ότι ο πολίτης ανησυχεί ιδιαίτερα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, αλλά δεν έχουμε να κάνουμε με την αποτροπή κλασικών εγκληματικών δομών και οργανώσεων, οργανωμένου εγκλήματος στον χώρο των ναρκωτικών, του λαθρεμπορίου ανθρώπων και τις νέες προσεγγίσεις και μορφές επίθεσης μπορούν να αξιοποιήσουν. Η πρόταση της οδηγίας αναφέρει για κάθε κράτος μέλος τον προσδιορισμό μιας αρμόδιας αρχής και διασύνδεση των δομών στο, στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας θα έχουμε τις υποδομές αυτές οι οποίες έχουν απόλυτη σημασία σε περίπτωση μιας κυβερνοεπίθεσης υπάρχει μια διαβάθμιση δηλαδή των δομών και των υπηρεσιών εκείνων οι οποίες είναι απαραίτητες για τη διαφύλαξη της ευημερία και εκείνων που δεν είναι τόσο απαραίτητες και έτσι θα πρέπει να προστατεύονται αυτές από ε, επιθέσεις. Και αυτό με είτε επίσημες είτε μη επίσημες ε, καταγγελίες ή αναφορές για επιθέσεις. Εκείνοι οι οποίοι βρίσκονται σε ιδιαίτερα ευνοϊκή θέση και μπορούν να γνωρίζουν καλύτερα και να αξιολογούν καλύτερα τους πιθανούς ή ε, επίκαιρους κινδύνους θα έχουν ιδιαίτερο ρόλο να διαδραματίσουν. Οι ε, έρευνες διοκτικές δραστηριότητες εν γέννη στα κράτη-μέλη θα σημαίνουν συμμετοχή ε, ε, ενός, ή προσδιορισμό ενός ενιαίου point of contact, σημείου επαφής, ώστε να μην, ε, να μην χάνεται η εστίαση με τη, λόγω της συμμετοχής πολλαπλών ε, υπηρεσιών και αρμοδίων. Η συνεργασία, όπως είπαμε, έχει πολύ μεγάλη σημασία και καλεί και τον συμμετέχοντα στην ε, δραστηριότητα, στην αγορά δηλαδή, να συμμετέχει δραστήρια, να ενημερώνει. Βέβαια η οδηγία πρέπει να είναι διατυπωμένη με τρόπο σαφή ως προς τον, τους τομείς οι οποίοι έχουν να διδραματίσουν τέτοιο ρόλο, Φερρυπίν αγορά ενέργειας, φερρυπίν συστήματα μεταφορών. Τομείς που όμως δεν σημαίνουν ότι κάθε επιχείρηση φέρει την ίδια ευθύνη ή ευθύνη στον ίδιο βαθμό. Μια ε, επιχείρηση η οποία διαχειρίζεται διευρωπαϊκά δίκτυα έχει πολύ μεγαλύτερες ευθύνες από μια ε, επιχείρηση διαχείρισης απο μια επιχειρηση διαχειρισης φωτοβολταικων ηλεκτρικών συστημάτων που εξυπηρετεί 300 σπίτια. Επισόδια λοιπόν ε, οι προβλήματα τα οποία μπορούν ε, να καταγράψουν μέσα σε ένα έτος οι αρχές αυτές και τα σημεία επαφή, μπορούν να δημοσιεύονται μια φορά το χρόνο σε μια έκθεση ώστε να γνωρίζει και ο πολίτης ε, ότι τα δίκτυα τα οποία χρησιμοποιεί από την άνεση του σαλονιού του μπορούν να είναι ευάλωτα, μπορούν να κινδυνεύουν από επιθέσεις. Με την οδηγία προσπαθούμε να προχωρήσουμε λίγο ακόμα στην ευαισθητοποίηση των πολιτών. Και θα αναφερθώ σε κάτι ακόμη. Η ασφάλεια και η καταγραφή ε, προσβολών αυτής έχει μεγάλη σημασία σε τομείς που έχουν πάρει διαστάσεις σημαντικές για την αγορά και πρέπει να γίνεται και αξιολόγηση από τον πάροχο της, ε, του πόσο ευάλωτα είναι τα συστήματά του, γιατί ο πάροχος είναι σε θέση να αξιολογήσει, πιστεύω ουσιαστικά, είτε ο ίδιος είτε με ανάθεση σε κάποιο τρίτο, ε, την ασφάλεια των συστημάτων του και θα μπορούσαμε, χωρίς βέβαια να επιβάλλουμε μια ενιαία ρύθμιση, η οποία θα ήταν και δύσκολο να εφαρμοστεί, αλλά και γραφειοκρατική υπερβολικά, να καλέσουμε τους παρόχους, αναλαμβάνοντας και τις σχετικές αρχές, αναλαμβάνοντας και τις, και τις δικές τους αρμοδιότητες ο καθένας, να μεριμνούν για την ασφάλεια των δικτύων. Στόχος επίσης και κατά την υλοποίηση της πρέπει ιδιαίτερα να προσέξουμε, είναι η διαχείριση του κινδύνου μέσα στις υποδομές της ίδιας, χωρίς επιβαρύνση γραφειοκρατική, η διαχείριση των πληροφοριών έχει σημασία. Και βέβαια στο μέτρο και στο μέγεθος των ε, φορέων της αγοράς. Ευελιξία λοιπόν είναι το κύριο αίτημα όσον αφορά τις ε, απαιτήσεις για ασφάλεια που θα επιβαρύνει τον κάθε παράγοντα ή φορέα της αγοράς η μη τήρηση των ε, ε, προϋποθέσεων τώρα ή των όρων αυτής της οδηγίας θα σήμαινε κυρώσεις ή όχι. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει κάποια διασύνδεση με κυρώσεις για να γνωρίζει ο παράγων, ο φορέας, ο πάροχος ότι υπάρχουν συνέπειες από την μη τήρηση των ε, υποχρεώσεών του. Και βέβαια στον τομέα του public policy, του δημοσίου δικαίου ουσιαστικά, δεν, μπορούμε να, δεν έχει νόημα να επιβάλλουμε κάποια διάταξη αν δεν τη συνοδεύουμε και κυρώσει. Γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ ουσιαστικό, πολύ σημαντικό και με τις τροπολογίες που προτείνω προς τους συναδέλφους νομίζω ότι βελτιώνεται ακόμη περισσότερο το κείμενο. Είναι ένα κείμενο στο οποίο εμπλέκεται και η Επιτροπή Βιομηχανίας και η Επιτροπή το... για τις Πολιτικές Ελευθερίες ε, Περιμένω να ακούσω φυσικά με πολύ ενδιαφέρον τι έχουν να πούν οι συνάδελφοι, αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Good. Well, thank you very much. Um, now, who else wants... Ευχαριστώ πολύ. Σμιτ Ρίλε, θέλετε να πείτε κάτι? Ε, to be honest. Ε, Ρίλε, για να είμαι ειλικρινής, είχε ο εισηγητής ο Σκιός από την ομάδα μας, ε, μου είχε δώσει μια γραπτή ε, δήλωση, αλλά αφού δεν υπάρχει κανεί σκιώδη, θα σας τη δώσω ή θα σα. Ε, εσάς ή στου συναδέλφου. Σμιτ. Και εγώ τον κύριο Μάντα αντικαθιστώ, που είναι άρρωστος. Και εγώ έχω μια γραπτή δήλωση. Τι να κάνω, τη διαβάσω ή να σας τη δώσω κι αυτή. Είναι καλή, πολύ καλή είναι, αλλά να σας τη δώσω κι εγώ, να μην τη διαβάσω. so, um, so I think we'll... Ωραία. Άρα ε, έχουμε μια ωραία ανταλλαγή γραπτών ε, δηλώσεων. Μπορεί βέβαια να τα διαβάσει ο κύριος ε, Σβάμπ, ε, όσο μιλάει ο κύριος Αλμόντι, και να μας πει τι λένε περιληπτικά. Εγώ τώρα όμως, ως και θέλω να σας πω εν συντομία ότι Πιστεύω ότι η γενική προσέγγιση που ακολούθησε ο κύριος Βάμπα ε, είναι μια προσέγγιση που με βρίσκει σύμφωνο. Ουσιαστικά ε, όταν είχε έρθει και ο εκπρόσωπο Κομισιόν να μας παρουσιάσει ε, τα σχετικά είχαμε και τη μελέτη αντικτύπου, είχα κάνει κάποια σχόλια. Πρέπει να λάβουμε δράση, το είπατε και εσείς, είναι σημαντικές πολιτικές δράσεις που πρέπει να γίνουν. Από την άλλη πλευρά η οδηγία αυτή νομίζω ότι είναι και φιλόδοξη σε σχέση με το τι πρέπει να γίνει στο παρόν στάδιο και νομίζω ότι ε, θα έπρεπε να μην παραγνωρίζει τις προσπάθειες των κρατών μελών που έχουν ή δεν έχουν ακόμη τις ε, ε, δομές αναφοράς. Έχουν γίνει πράγματα στα κράτη μελή. Τώρα σε ό,τι αφορά την υποχρεωτική υποβολή αναφορών, ε, δεν ξέρω αν θα συμφωνούσα. Νομίζω ότι είναι ένα πρόβλημα για τις επιχειρήσεις. Η υποχρεωτική υποβολή αναφορών σε κάποιες περιστάσεις θα μπορούσε να αποτρέψει τις επιχειρήσεις από το να σχεδιάσουν την ασφάλεια και να αναζητούν παραβάσεις, παραβιάσεις αυτής. Εξορισμού, όταν μιλάμε για υποχρεωτική υποβολή αναφορά, ότι κάποιος πρέπει να λάβει εντολή να συντάσσει αυτές τις εκθέσεις και να τις λαμβάνει. Φοβάμαι ότι θα μπουν πολύ στον πειρασμό να συμπληρώνουν, να τσεκάρουν τετραγωνίδια και να στέλνουν την έκθεση έτσι. Αλλά τα θέματα αυτά είναι σημαντικά και νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει μια αλλαγή συμπεριφορά. Αυτό είναι ο στόχο τη Κομισιόν, δεν απατώμε. Πώ όμω με μια νέα δομή απλά πετυχαίνει κανεί αλλαγή συμπεριφορά και με την ε, κυκλοφορία κάποιων εγγράφων ε, στα οποία έχουν απλά τσεκαριστεί κάποια τετραγωνίδια. Ε, δείχνει σίγουρα όλο αυτό ότι υπάρχουν κάποιες ανεπάρκειες και ότι πρέπει να είμαστε πιο ρεαλιστές. Δεν είναι μόνο δική μου προσέγγιση, νομίζω ότι συμφωνούν αρκετοί με αυτό. Και σε ό,τι αφορά τις ε, απαιτήσει για την υπόβλη αναφορών πρέπει να είναι πραγματιστικές. Ποιος θα διαβάσει τις αναφορές αυτές Πρέπει να έχουμε πραγματικούς στόχους. Εγώ συμφωνώ με το ότι η Επιτροπή μας, με το Συμβούλιο, ακολούθησε μία προσέγγιση για τις απαιτήσεις κοινοποίηση. και σε μια άλλη περίπτωση. Και σε ό,τι αφορά τα δεδομένα και την προστασία των δεδομένων, πάλι έπρεπε να οριστούν τα δεδομένα και οι παραβιάσεις αυτής της εμπιστευτικότητας. Πρέπει λοιπόν να είναι πολύ σαφείς οι περιγραφές για τις παραβιάσεις που είναι σημαντικές, γιατί έχουν και συγκεκριμένες επιπτώσεις. Μια τέτοια προσέγγιση θεωρώ ότι πρέπει να εφαρμοστεί και στην προκειμένη περίπτωση και είμαι απογοητευμένος γιατί το έργο ε, που έχει γίνει σε ό,τι αφορά την προστασία δεδομένων, για παράδειγμα, δεν το έλαβε υπόψη της η Κομισιόν. Κάποιος ιός φαίνεται να υπάρχει στην Κομισιόν αυτή τη στιγμή, δηλαδή ε, μανία να στέλνουμε εκθέσεις μακροσκελέστατες, να ανταλλάσσουμε κείμενα, μα τελικά έτσι δεν κάνουμε τίποτα στην πράξη. το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών δεν είναι ικανοποιητικό, πρέπει να το δούμε. Ο Ανδρέας, νομίζω με τροπολογία 9, προς τα εκεί κινείται κάπου. Απλά θα τον ενθάρρυνα να επαγρυπνήσει περισσότερο προς αυτό το θέμα, γιατί χρειαζόμαστε και μεγαλύτερη ευελιξία σε θέματα ανταγωνισμού και διακριτική ευχαίρεια που θα πρέπει να έχουν οι αρχές. Διότι πρέπει να έχουμε υπόψη μα ότι στα 25, στα 28 συγγνώμη, κράτη-μέλη τη Ένωση υπάρχουν τεράστιε διαφορέ ό,τι αφορά τι δυνατότητε και ικανότητε αντιμετώπιση αυτών των ε, ζητημάτων. Και κάθε τέτοιου είδου νομοθεσία, κατά την άποψή μου, θα πρέπει να μπορεί να λάβει αυτό το στοιχείο υπόψη. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν ε, πρέπει να επαγρυπνούμε, γιατί θα μπορούσε μια παραβίαση να συμβεί το ίδιο εύκολα σε μια μεγάλη όσο και σε μια μικρή χώρα. Και υπάρχει τάση βέβαια να στοχεύονται οι πιο, οι πιο αδύναμες ε, χώρες, αλλά τα προληπτικά μέτρα είναι αυτά που θα πρέπει να ε, μας απασχολήσουν καταρχήν, πιστεύω. Δεν είναι ο σωστός τρόπος κατά ανάγκη να δημιουργήσουμε νέες δυσκίνητες γραφειοκρατικές δομές. Ο Αντρέας λοιπόν νομίζω πως τη σωστή κατεύθυνση κινείται με τις προτάσεις του, ως σκιώδης σε αυτό διαπιστώνω. Λοιπόν, αυτά να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Κομισιόν για να μας πει και αυτός αρχικά τι πιστεύει για την έκθεση ΣΒΑΠ. Um, thank you very much and good afternoon. Ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον Αντρέα Σουβάμπ, πολύ καλή έκθεσή του. Και πάλι ε, διαφαίνεται ότι κατανοεί τις ε, ανησυχίες μας καθώς και τις ανάγκες που υπάρχουν για την οδηγία ε, και είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος, η και η Επιτροπή, σε μεγάλο βαθμό. Αυτά τα περιστατικά σε σχέση με την ασφάλεια σχετίζονται με την εθνική ασφάλεια. Δεν πρέπει να μπερδευόμαστε. Σωστά το είπε ο εισηγητής. Η οδηγία αυτή σχετίζεται με την ευημερία, την ανάπτυξη, την απασχόληση και ουσιαστικά ε, την ε, διαφύλαξη της εσωτερικής αγοράς ε, ενισχύοντας την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα των συστημάτων ασφαλείας που στηρίζουν βασικές οικονομικές και κοινωνικές διαδικασίες που είναι και στη βάση της λειτουργίας της ψηφιακής αγοράς. Θα είμαι όσο πιο σύντομος γίνεται τέσσερα σημεία είναι βασικά και σχετίζονται με την έκθεση ε, του κυρίου Σφάμπ. Ποια είναι τα σημαντικά σημεία για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχουμε πάνω από μία αρμόδιες εθνικές αρχές. Ε, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα Ε, αναφέρεται εξάλλου και στην έκθεση υπάρχει μία μονοστάση για την ε, συνεργασία ως προς την ανταλλαγή πληροφοριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, δεύτερον, το πεδίο εφαρμογής ε, για τις υποχρεώσεις υποβολής αναφορών για την ασφάλεια στο άρθρο 14 της πρότασης. Αυτές οι υποχρεωτικές απαιτήσεις υποβολής αναφοράς ε, είναι κάτι πολύ σημαντικό για μας. Σε κάποια κράτη-μέλη υπάρχει ε, θελούσια συνεργασία και μπορεί όντως να έχει αποτελέσματα. Όμως, σε άλλες περιπτώσεις, ε, η συνεργασία ανάμεσα στους οικονομικούς φορείς και τις αρμόδιες εθνικές αρχές, όταν υπάρχει, δεν λειτουργεί αισίως ή είναι ανύπαρκτη, όπως σας έλεγα. Γι' αυτό επιμένουμε για αυτές τις υποχρεώσεις υποβολής αναφορών ε, για τα περιστατικά και για τη διαχείριση του κινδύνου. Χρειαζόμαστε αυτά τα στοιχεία για την εκπόνηση των εθνικών στρατηγικών και για την αρρωγή των οικονομικών φορέων που έχουν βιώσει ένα τέτοιο περιστατικό και ε, για να περιορίσουμε τις αρνητικές συνέπειες χρησιμοποιώντας το εθνικό σύστημα ε, ασφαλείας. Ε, αυτό το χρειαζόμαστε για τους βασικούς προμηθευτές υπηρεσιών. Ε, ως προς το, τις βασικές διατάξεις αντιλαμβάνομαι όντως ότι είναι υπερβολικά φιλόδοξη η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όμως είναι πλήρως δικαιολογημένη αυτή η φιλοδοξία που έχουμε. Οι πύλες ε, για τις ηλεκτρονικές ε, πληρωμές, ε, για τις ηλεκτρονικές αγορές, τα ηλεκτρονικά καταστήματα για τις ψηφιακές εφαρμογές μπορούν να θεωρηθούν ως βασικοί παίκτες της αγοράς γιατί σε αυτούς φορείς αντιστοιχεί μεγάλο ποσοστό ηλεκτρονικών συναλλαγών και υπάρχουν πολλά οικονομικά στοιχεία των χρηστών, των αγοραστών. Οπότε θεωρούνται βασικοί παίκτες γιατί είναι σημαντικά αυτά τα στοιχεία και για τη συνέχεια των εμπορικών συναλλαγών, ε, των ηλεκτρονικών συναλλαγών ε, και ε, ε, μια βασική παρενέργεια, αν θέλετε, της οδηγίας είναι και η τύχη των οικονομικών δεδομένων που χρησιμοποιούνται για τις επιγραμμικές συναλλαγές. Αν περάσουμε τώρα στα δίκτυα, μπορούμε να κάνουμε ένα παραλληλισμό με τα δίκτυα, τα ηλεκτρονικά δίκτυα ε, επικοινωνίας. Αυτά τα κοινωνικά δίκτυα ε, πλέον έχουν γίνει επικοινωνιακοί κόμβοι που παρισφρίουν παντού, ε, είναι πανταχού παρόντα και απαραίτητα κιόλας για την συνδεσιμότητα της Ευρώπης. Ε, εμένα δεν θα με εξέπλητε αν σε λίγα χρόνια η Ευρώπη υπηρεσίε όπως το Twitter ή το Facebook ε, έχουν ακόμη ε, μεγαλύτερη βαρύτητα ως προς την συνδεσιμότητα κατά τη διαστολή, δηλαδή με παραδοσιακούς τηλεπικοινωνιακούς φορείς για την αναλογικότητα και το είδος των ε, περιστατικών ασφαλείας που πρέπει να αναφέρονται. Τι κάναμε αντιγράψαμε το άρθρο 13α της ε, Οδηγίας Πλαίσιο για τις Τηλεπικοινωνίες. Εάν κρίνεται, όπως πιστεύει ο εισηγητής, ότι θα έπρεπε να εξηγήσουμε καλύτερα και να παραθέσουμε τις περιστάσεις υπό τις οποίες ένα τέτοιο περιστατικό επηρεάζει τους βασικούς ε, Παρόχου ε, υπηρεσιών και του βασικού παίκτε τη αγοράς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι στην πρόταση γιατί έτσι μπορεί να ενισχύσουμε ε, και την νομική ασφάλεια. Συμφωνούμε και πάλι λοιπόν με τον εισηγητή και τέλο. Ένα δευτερόλεπτο και θα κλείσω για το θέμα της ευθύνης. Πιστεύουμε ότι είναι καλό που συμπεριλαμβάνεται αυτό στο πεδίο οδηγία. Ένα ε, Ένας ε, φορέ ε, κρίσιμη υποδομή ή οποιοδήποτε ο οικονομικός φορέας μπορεί να υποφεληθεί, διότι αν εκείνος μπορεί να εξασφαλίσει ότι θα συμμορφωθεί με τους κανόνες, εν τη αυτή περιπτώσει είναι εύκολο να έχουμε ένα τεκμήριο της ε, δέουσας επιμέλειας για τον οικονομικό φορέα εν τη αυτή περιπτώσει. Δεν φέρει η αντίποτε αστική ή ποινική ευθύνη σε περίπτωση δίωξη αυτός ο οικονομικός φορέας. Αυτό μπορούμε να το φτιάξουμε μαζί. Δηλαδή, ξαναλέω, τεκμήριο επαγγελματικής επιμέλειας για τον οικονομικό φορέα. αν σε περίπτωση που εντάσσεται στο πεδίο εφαρμογή αυτός ο οικονομικός φορέας και συμμορφώνεται όμως και με τι απαιτήσει υποβολής αναφόρων. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ Ξεκάθαρε οι απαντήσεις σας. Αντρέα, θέλεις ε, ε, να κάνεις κάποιες ε, καταληκτικές παρατηρήσεις και ενδεχομένως να μιλήσει για την αλλαγή του χρονοδιαγράμματος. Έχω φτιάξει ένα λογίδρο για τα υπόλοιπα 24 λεπτά. Πρώτα απ' όλα. Θα ήθελα να συμφωνήσω και εγώ με αυτή την προσέγγιση και με τις ερωτήσεις που θέσατε κι εσείς όταν ε, ε, μιλήσατε. Ευχαριστώ τον Ματία Έγκστρομ που συνέταξε αυτά τα σχόλια και να ευχαριστήσω και τον Όλε Σμιτ και την κυρία Λολίν που μου έδωσαν αυτές τις παρατηρήσεις. Ο κύριος Μέντες μου γράφει εδώ ότι συμφωνεί με αυτά που λέω, αλλά επιθυμεί μια εξαίρεση για τις μικρές επιχειρήσεις από δυσανάλογα βαριές υποχρεώσεις. Κατά τη γνώμη μου δεν είναι δυσανάλογα βαριές, αλλά και εγώ ίδιος Πρότεινα ούτως ή άλλως οι μικροεπιχειρήσεις και μικρές επιχειρήσεις να εξαιρεθούν. Για τις μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις μάλλον θα αποδειχθεί αυτό δύσκολο. Ο κύριος Έγκστρομ έδωσε μια ευρύτερη εξήγηση. Προτείνει τη σύσταση και όχι την οδηγία γιατί για την κυβερνοασφάλεια κρίνω τα κράτη-μέλη δεν αρμόδια να δίνουν ε, την κατεύθυνση. Υπό το φω ε, τη ε, περαίουσα πολιτική ατμόσφαιρα, και εγώ το θεωρώ κοπλιμέντο, δεν θεωρώ την κριτική από πλευρά του, ότι η οδηγία είναι το πλέον αποδεκτό εργαλείο και καλωσορίζω τι τροπολογίε του εισηγητή προ αυτή την κατεύθυνση. Λοιπόν, θα συμφωνήσω με αυτή την τοποθέτηση και χαίρομαι επίση, διότι ο Τζουζέπε με τον οποίο συνεργαστήκαμε για την οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών ε, στην αρχή της θητείας μας έκανε πάρα πολύ κέρια σχόλια και θέλω να επανέλθω σε αυτά. Λοιπόν, η οδηγία, ε, αν, συμπεριληφθούν, αν ληφθούν υπόψη οι τροπολογίες μου, τι σημαίνει ότι η πάροχη σε τομείς ε, κέριων υποδομών που έχουν εκτιμήσει ότι αντιμετωπίζει κρίσιμη κατάσταση κυβερνοεπίθεσης η κέρια αυτή η υποδομή πρέπει να αναφέρουν το περιστατικό μόνο όταν είναι, και λέμε στα αγγλικά, of significant importance, αρκετά σημαντικό. Τι κάνουμε, Περιορίζουμε το πεδίο εφαρμογή, ε, διότι για τι κέρυε υποδομέ έχουμε βγάλει ήδη δύο κατηγορίε που είχε συμπεριλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και παρενθετικά να πω ότι μπορούμε να το συζητήσουμε αν είναι ε, η καλύτερη οδό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, συρρυκνώνεται σημαντικά το πεδίο εφαρμογή και λόγω αυτού δεν είναι αρκετά υψηλέ οι απαιτήσει υποβολή αναφορών. Για να είναι όμω λογικά αυτά, θα πρέπει να προβλέπεται μια ε, υποχρέωση αναφορά τέτοιων σημαντικών περιστατικών. Ουδάλλως δεν θα λειτουργήσει το δεύτερο σημείο. Ε, η δημόσια διοίκηση δεν εμπίπτει σε αυτό το πεδίο εφαρμογή. Εγώ πιστεύω ότι εκφύσεως ε, ε, θα προστατεύσουν τις κύριε υποδομές και άρα θα υποβάλουν αναφορά. Όταν εν μέρει έχουν ιδιωτικοποιηθεί αυτές οι υπηρεσίες, μπορεί να συμπεριληφθούν στην οδηγία ούτω ή άλλως, Προ το παρόν όχι. Και ούτω ή άλλω αυτό θα είναι συνάρτηση του κατά πόσο αυτή η κρίσιμη υποδομή ε, ανήκει στην κατηγορία των υποδομών που ε, ενδέχεται να δεχτούν τέτοιες κυβερνοεπιθέσεις. Ε, όπου υπάρχουν αντιρρήσεις ε, μπορούμε ενδεχομένως να επεξεργαστούμε αυτά τα σημεία. Κάποιοι θα ήθελαν να απορρίψουν τελείως την ιδέα της οδηγίας, όμως λόγω του πολιτικού κλίματος που επικρατεί, όπως λέει ο κύριος Έγκστρομ, δεν μπορεί το Κοινοβούλιο να πει «Α, όχι, δεν θα κάνουμε τίποτα γιατί είναι δύσκολο να το καταφέρουμε». Όχι, πρέπει κάτι να κάνουμε για να συνειδητοποιήσουν οι πολίτες ότι φέρουν και οι ίδιοι ευθύνε, γιατί σε αυτό δεν αναφερόμαστε και αυτές οι υποδομές που πραγματικά είναι κρίσιμη σημασία για την καθημερινότητα των πολιτών θα εμπέσουν στο πεδίο ε, εφαρμογής οδηγίας. Τον περασμένο μήνα έκανα πολλέ. Ε, επαφές για τον ορισμό. Τι σημαίνει κρίσιμη υποδομή. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Κάποιοι μου είπαν ότι και τα ΜΜΕ πρέπει να συμπεριληφθούν γιατί όταν υπάρχει κρίση οι άνθρωποι πρέπει να έχουν πρόσβαση στο BBC ξέρω εγώ. Αν δεν λειτουργεί το BBC μπορούν να πάνε στο CNN ή σε άλλα ΜΜΕ. Και μπορούμε να δούμε από αυτό το παράδειγμα ότι οι πολίτες πάντοτε έχουν άλλες επιλογές. Αυτή οι τομή που αναφέρονται στο πεδίο εφαρμογής είναι όντως κρίσιμη σημασία και όντως πρέπει να μεριμνούμε για την ασφάλειά τους. Την επόμενη φορά ε, μπορούμε να εξετάσουμε τροπολογίες που ενδεχομένως να κατατεθούν. Τώρα 24 Σεπτεμβρίου θα γίνει αυτό, 1η Οκτωβρίου θα είναι καταληκτική ημερομηνία για τις, ε, την υποβολή τροπολογίων, δεν ξέρω, αποφασίστε το εσείς Πρόεδρε, αλλά νομίζω ότι ε, καλύτερα να σπεύσουμε παρά να περιμένουμε. Την ε, Τον Ιούνιο πήραμε την πρόταση αυτή Οπότε είχαν χρόνο να τη συζητήσουν και να τη διαβάσουν οι συνάδελφοι ε, και ευελπιστούμε, αν συμφωνήσει και η Επιτροπή, να επιδιώξουμε την πρώτη, τη συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση. Προσβλέπω στις μελλοντικές συζητήσεις και σας ευχαριστώ για την αμύωτη προσοχή σας. Ε, Πρόεδρος, 24 Σεπτεμβρίου. Καλό μου φαίνεται. Γιατί χρειαζόμαστε οπωσδήποτε τη συμβολή της Επιτροπής Βιομηχανίας. Ε, πρέπει να έρθετε σε επαφή με την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, αν υποθέσουμε ότι έχουν εισηγητή και ότι είναι έτοιμοι, να του πείτε ότι πρέπει να βιαστούν. Γιατί με την οδηγία προστασία των δεδομένων ε, στο πολιτικό ζήτημα σημειώθηκαν μεγάλε καθυστερήσει και είναι απαράδεκτο. Δεν μπορεί να επαναληφθεί. Πρέπει να βιαστούμε για την ε, οδηγία για τα προσωπικά δεδομένα έχουν καθυστερήσει τόσο πολύ που δεν κάνουν πια τίποτα. Μπορεί να βρουν χρόνο να ψηφίσουν για αυτό. Δεν ξέρω το αν υπερβολικό από πλευρά μα να του το ζητήσουμε, αλλά τέλο πάντων. Αν θέλετε βοήθεια από πλευρά μου για να τα συζητήσετε με τον Πρόεδρο και τον εισηγητή, ευχαρίστω. Και για την Επιτροπή τι θα πω, θέλω να αρχίσουμε το συντομότερο δυνατόν τις συζητήσεις ε, με το Συμβούλιο, αλλά όπως καταλαβαίνετε πρέπει πρώτα να περάσει το θέμα από την ε, διάσκεψη των Προέδρων. Ε, Αντρέα, ευχαριστώ για τον ηγετικό σου ρόλο και τις προσπάθειες. ευχαριστώ όλους τους παρισταμένους ε, ολοκληρώνει τη συνεδρίαση και στις 25 Σεπτεμβρίου την Τετάρτη από τις 9 μέχρι τις 6.30 και την 5η 26 Σεπτεμβρίου από τις 9 μέχρι τις 6.30. Επίσης, ε, γιατί τότε είναι και η ψηφοφορία στις 10 το πρωί, θα γίνει η επόμενη συνεδρίασή μας, θα τα πούμε τότε. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας σήμερα το απόγευμα, όσοι ήσασταν ακόμη εδώ πέρα και καλό βράδυ.